Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ να πάρουμε τις θέσεις μας. Βεβαίως μετά την συνεδρίωση των ιστών δεν είχαμε και πολύ χρόνο για το διάλειμμα, για το γεύμα, αλλά ε, είναι περασμένες τρεις και πρέπει να επανέλθουμε στις εργασίες μας. Προχωρούμε λοιπόν και να χαιρετήσουμε, να καλωσορίσουμε βεβαίως την Επίτροπο Αρμόδια για θέματα ιστορικών υποθέσεων, την κυρία Σεσίλια Μάλνστρομ. Σας καλωσορίζουμε εκ νέου, κυρία Επίτροπε. Είναι τιμή μας να σας έχουμε μαζί μας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2012 και τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε ό,τι αφορά το σύστημα εισόδου-εξόδου, την ανομική βάση για τη Europol και την επανεξέταση της οδηγίας για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, γενικότερα οι προτεραιότητες ε, για το 2012 υψηλούν ενδιαφέροντος για την Επιτροπή μας θα ακούσουμε τι έχει να μας πει η Επίτροπος και μετά θα δώσουμε το λόγο στα μέλη για συζήτηση. Η κυρία Μάλστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Προσβλέπω σε μια καλή χρονιά και συνεργασία μαζί σας να συγχαρώ για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Ήδη είστε στο της θητείας σας. Οπότε είναι καλή η ευκαιρία, μια και εμεί είμαστε εμεί τη θητεία μα στην Επιτροπή, να ε, κάνουμε έναν απολογισμό των πεπραγμένων και τι έχουμε μπροστά μα. Η περσινή χρονιά ήταν μια καλή χρονιά σε επίπεδο συνεργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου καθώς ε, απέδειξε, το αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει συνεργασία Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Βεβαίως, η περσινή χρονιά ήταν δραματική, η οικονομική κρίση συνεχίζει να υπάρχει και όλα, όλες οι πολιτικές επηρεάζονται και οι πολιτικές που απασχολούν εσάς επηρεάζονται. Και βεβαίω το θέμα της οικονομικής κρίσης είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οπότε ίσως... Ε, είναι και καλό το ότι και εμεί εργαζόμαστε επί θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερου πολίτε μα. Βεβαίω αυτό σημαίνει και πολύ μεγάλη ευθύνη για όλου μα. Πριν τα Χριστούγεννα, πριν διακόψουμε για τα Χριστούγεννα, είχαμε μια πολύ στενή ε, συνεργασία ανάμεσα στην για να υιοθετηθεί η πρόταση για την ενιαία άδεια, εξαιρετική πρωτοβουλία για να διευκολύνουμε τη ζωή των μεταναστών με την ε, επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και την ε, διασφάλιση της ίσης ε, μεταχείρισης. Επίσης, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί εθετήθηκε και η οδηγία για τις προϋποθέσεις και ήταν πραγματικά πολύ σύνθετες, δύσκολες προτάσεις στα πλαίσια του συνολικού πακέτου για το άσυλο. ευχαριστώ για την σχετική προσπάθεια το φθινόπωρο, αλλά ακόμη και τώρα κυρίως αυτό που με απασχολεί είναι το follow-up για, το πακέτο του Σέγγεν θα επανέλθω σε αυτό το θέμα σε λίγο. Επίσης να πω ότι η οδηγία για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας έχει υιοθετηθεί και έτσι μπορούμε να προσθέσουμε καλύτερα τα παιδιά μας. Επίσης, υιοθετήσαμε τον εξυγχρονισμένο κανονισμό για τα πυροβόλα όπλα. Επίσης, έχουμε τη νέα εντολή για την Frontex για να ενισχυθεί η ο επιχειρησιακό χαρακτήρα τη Frontex, αλλά και έτσι να ενισχύσουμε και το χάρτη των δικαιωμάτων μέσα από αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε, λοιπόν, και μετά το πρώτο έτο αξιολογήσεων ε, των σχεδίων δράση για την ασφάλεια να έχουμε να... μια καλή εικόνα τη κατάσταση λοιπόν ένα χρόνο μετά. Έπειτα, ο αγώνα κατά της τρομοκρατία και του εγκλήματο. Έχουμε προχωρήσει και εκεί, ολοκληρώσαμε τι διαπραγματεύσει και ε, τη συμφωνία PNR με την Αυστραλία, από ό,τι θα γνωρίζετε. Μονογραφήσαμε την ε, συμφωνία PNR με τις Πολιτείες που αυτή τη στιγμή εξετάζετε εσείς και έχουμε επιτύχει και σημαντική πρόοδο στις προτάσεις ε, σχετικά με τη χρηματοδότηση όλων των πολιτικών εσωτερικών υποθέσεων. Ήταν πραγματικά πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμα το φθινόπωρο που αφορούν τους νότιους γειτονές μας και το όλο πακέτο για τη μετανάστευση είναι κάτι που θα μας συνεχίσει να μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα. Τώρα, από εδώ και πέρα, μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες για το υπόλοιπο θητείας μας είναι το κοινό ε, σύστημα ασύλου. Είναι κάτι που συζητήσατε και το πρωί με τον Οδανό Υπουργό, ο οποίο έχει δεσμευτεί να προωθεί σε αυτό το φάκελο και εγώ είμαι απόλυτα δεσμευμένη να συνεργαστώ μαζί σας, όπως φαίνεται ίδιο τώρα και με τους εισηγητές και τους σκιώδες εισηγητές να προχωρήσουμε ώστε να έχουμε μια καλή συμφωνία τελικά για όλο το πακέτο. Η συμφωνία στο Συμβούλιο για την Επανεγκατάσταση είναι πολύ καλό μήνυμα προς αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζω ε, και εμεί και η Ιδανική Προεδρία να προχωρήσει συζητήσει για τις συνθήκες υποδοχής να έχουμε τριμερεί διαλόγου στο σημότερο δυνατόν για να προχωρήσουμε και αυτό το θέμα. Αυτό βεβαίω συνδέεται και με την οδηγία για τι διαδικασίε. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά και για του δύο φακέλου θα πρέπει να επιτύχουμε πρόοδο. Όσον αφορά το κανονισμό του Δουβλίνου, αυτό ξέρω ότι είναι ακανθόθε ζήτημα και ξέρω ότι το παρακολουθείτε με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε ξεκινήσει μια ευρύτατη συζήτηση και για ένα μηχανισμό και ένα ε, μηχανισμό εγκύρης προειδοποίησης για τον ε, αξιολόγηση ε, του κανονισμού του Δουβλίνου. Χρειαζόμαστε όμως ένα μηχανισμό που να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να έχουμε καλούς κανόνες εύκολα εφαρμόσιμους. Μπορούμε να δουλέψουμε πολύ καλά μόνο αν αυτό συνοδευτεί και από πραγματικά μέτρα Επίτα. Σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς μετανάστες, ε, θα πρέπει να επιτύχουμε πρόοδο και εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να επιτύχουμε πρόοδο και σε ό,τι αφορά την ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση και τη σχετική οδηγία πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσει μεταξύ των οργάνων για αυτό το ζήτημα. Εκτιμώ τη δική σα προσπάθεια για την ενίσχυση ε, του δελεαστικού χαρακτήρα αυτού του προγράμματο του ενδοεπιχειρησιακή ε, μετάθεση. Έπειτα, εκτιμώ τη θέση σα για του εποχικού εργαζόμενου και ελπίζουμε να υπάρξει σύντομα συμφωνία για αυτό το θέμα, ώστε να ανοίξουμε το δρόμο και για του υψηλά ε, και για του χαμηλά ειδικευμένου εργαζόμενου από τρίτε χώρε. Βεβαίω, οι μετανάστε έχουν δικαίωμα και στον οικογενειακό βίο γνωρίζω ότι μόλις χθες συζητήσατε ε, την πράσινη βίβλο που παρουσιάσαμε για την επανένωση οικογενειών. Προσβλέπουμε σε συνεργασία και σε αυτό το τομέα. Επίσης να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ισχυρή υποστήριξη που έχει δώσει το Ευρωκοινοβούλιο ε, όλες τις πολιτικές ομάδες στο πακέτο Σέγγεν. Ποτέ δεν έχετε ξεχάσει και εσείς τη σημασία του Σέγγεν για όλους τους πολίτες. Είναι μεγάλο επίτευμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Βεβαίως, Κατανοείτε ότι και εγώ αυτό το υπερασπίζομαι πολύ στεναρά. Βεβαίω, οι κανόνε έγκεν θα πρέπει να αναθεωρούνται όταν αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να προκαταλαμβάνουμε καλύτερα τα προβλήματα και να έχουμε ένα πιο ισχυρό μηχανισμό αξιολόγηση προ το συμφέρον των θεσμών και των πολιτών. Γιατί η διαχείριση των συνόρων και να μειώσουμε τη δυνατότητα, ε, μόνο τις περιπτώσεις όπου θα έχουμε την ad επαναφορά ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα. Επίσης, οι κανόνες που δεν έχουν εφαρμοστεί πολύ καλά να αντικατασταθούν από καλύτερους κανόνες. Είμαι πεισμένη ότι μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο και προσβλέπω να συνεργαστώ μαζί σας, όπως έγινε έως τώρα με τους κυρίους Κοέλιο και Βέμπε, εισηγητές ε, για αυτό το τόσο σημαντικό φάκελο η πολιτική θεωρήσεων σημαντική και για εσά και για μας και προωθούμε την πρόταση για την ε, ρήτρα διασφάλισης ώστε να υπάρχει προσωρινή αναστολή ε, της υποχρέωσης θεωρήσεων όποτε αυτό αγκαίο, Το Συμβούλιο ΔΕΗ πριν τα Χριστούγεννα συμφώνησε επί της γενικής προσέγγισης ώστε οι σχετικές αποφάσεις ε, να εξαρτώνται λιγότερο από αριθμητικά κριτήρια και γνωρίζω ότι και αυτή είναι και η δική σας προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αυτό το εργαλείο θα είναι μόνο η ίστατη λύση. Μόνο για έκτακτα πραγματικά γεγονότα. Συνεχίζουμε επίση του διαλόγου για περαιτέρω διευκόλυνση θεωρήσεων. Την περασμένη εβδομάδα μου στο Κωσυφοπέδιο και να ξεκινήσω διάλογο για τι θεωρήσει με την ε, κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου και περιμένουμε να πετύχουμε σχετική πρόοδο και με τι άλλε χώρε. Γενικότερα, θέλουμε να ενισχύσουμε το διάλογο με τις χώρες, τις τρίτες χώρες στη γειτονιά μας για την ενίσχυση των κανόνων μετανάστευσης και την ασφάλεια και αυτό είναι κομμάτι της σφαιρικής προσέγγισης που ε, ε, ανακοινώσαμε τον Νοέμβρη. Εταιρικέ σχέσει κινητικότητα. Ε, είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο με τρίτες χώρες στη γειτονιά μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο ε, στην γειτονιά μας, ε, στην Νότια Μεσόγειο. Είναι ένα γενικό σημαντικότερο ε, εργαλείο για να ενισχύσουμε την κινητικότητα τις ε, ατομικές ελευθερίες, αλλά από την άλλη να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στα σύνορά μας. Έχουμε συμφωνίες με την Ισία και το Μαρόκο και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και οι άλλες χώρες της περιοχής. Επίσης, μέσα στο 2012 θα σας παρουσιάσουμε και προτάσεις για τα έξυπνα σύνορα, για τη βελτίωση της ασφάλειας, αλλά και να διευκολύνουμε την, ε, τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν καλή την πίστη και πιστεύω ότι θα έχουμε και μια καλή συνεργασία και με αυτό το φάκελο ε, και σε, και με όλους εσάς. Έπειτα, πολέμηση της διαφθοράς. Ξέρω ότι υποστηρίζετε πάρα πολύ την ανακοίνωση της Επιτροπής και προσβλέπω συνεργασία και σε αυτό το τομέα μαζί σας. Γνωρίζετε ότι μόνο στα 27 κράτη-μέλη η Φυλακτική προσέγγιση είναι ότι 120 δις χάνουμε ετησίω λόγω διαφθορά. Και αυτέ είναι επιφυλακτικέ εκτιμήσει και δεν μιλούμε για διαφθορά που απορρέουν από σοβαρέ μορφέ εγκλήματο, ναρκωτικά κτλ. Κατανοείται λοιπόν πόσο σημαντική είναι η αιστεία σε αυτό το τομέα και αυτό θα προετοιμάσει και την έκθεση που θα εκπονήσουμε για του χρόνου. Ε, σε λίγε εβδομάδε επίση, και πάλι για το οργανωμένο έγκλημα θα υποβάλουμε προτάσει για το πώ μπορούμε να προστατεύσουμε την νόμιμη οικονομία από το οργανωμένο έγκλημα και να έχουμε καλύτερα εργαλεία για την ε, προσωρινή δέσμευση και δίμευση ε, των προϊόντων εγκλήματος. Τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα είναι πεπαλαιωμένα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, οπότε θα ε, περιμένετε τι νέε προτάσει τη Επιτροπή για τη δέσμευση και την κατάσχεση προσωπικών στοιχείων. για τα θέματα PNR βεβαίως, ε, ξέρετε την πρότασή μας, κοινή κανόνα στον τομέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, αρκεί να έχουμε υψηλά ε, πρότυπα προστασίας, ε, ασφάλειας, αλλά και διαφύλαξης των δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων. Το PNR με τις ΗΠΑ σας έχει υποβληθεί για έγκριση. Σα έχουμε στείλει την θέση της νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελπίζουμε να σας διευκολύνει κατά την δική σας αξιολόγηση της θέση σα. Πιστεύω ότι η συμφωνία που έχουμε ενώπιόν μα είναι μια εξαιρετική πρόοδο σε σχέση με την κείμενη συμφωνία, όπω και είναι τα σημαντικά βήματα που έγιναν από το Μάιο και μετά, απόδειξη αυτή τη συμφωνία. Επίση αντικατοπτρίζει ένα μήνυμα που αποστέλουν και τα τρία θεσμικά όργανα προ την Αμερικανική πλευρά. Χρειαζόμαστε πιο ισχυρέ διατάξει και μια πιο ε, συγκεκριμένη θέση από το θέμα. Έχουμε προόδο στη συζητήση με τον Καναδά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για αυτό το τομέα τώρα. Επίσης να αναφερθώ στο σύστημα εντοπισμού της χρηματοδότησης των υπάρχει πλέον ε, ένα κείμενο που εκπονούμε, υπάρχει μελέτη αντικτύπου που θα είναι έτοιμη την Άνοιξη, θα σας υποβάλουμε μια σχετική πρόταση και ελπίζουμε να προχωρήσουμε τη σχετική συζήτηση και με σας και με το Συμβούλιο σύντομα. Επίσης έχει αρχίσει η εξέταση οδηγίας αναθεώρησης τις οδηγίες για την διατηρήση προσωπικών δεδομένων Θεωρούμε ότι η νομοθεσία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για τι διοκτικέ αρχέ, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί σχετική νομοθεσία και εξετάζουμε ποιε είναι οι δυνατότητες, οι καλύτερες δυνατότητες επικαιροποίησης οδηγίας. Αυτά τα λέω για να σα ανοίξω λιγάκι την όρεξη, λέγοντά σας όμως ότι το, το Συμβούλιο δεν έχει καμία διάθεση για σημαντικέ αλλαγές. Ελπίζω το Κοινοβούλιο έχει μια άλλη στάση. Έπειτα, αργότερα την Άνοιξη, θα σα υποβάλουμε προτάσει για τη δημιουργία ενό κέντρου για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματο. για για να μπορούμε να ε, συντονίσουμε καλύτερα τις ομάδες αντίδρασης και να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματικό σύστημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ελπίζω η σχετική ανακοίνωση που θα έρθει την άνοιξη να μας βοηθήσει όλους για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Επίσης γνωρίζω ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό έγκλημα ε, είναι κάτι που ζητάτε κι εσείς και ελπίζω να συμφωνήσετε επί αυτού του φακέλου πριν το καλοκαίρι για τους υπολογιστές. Είχα τη δυνατότητα να πω και στον κύριο Κοέλιο πριν ότι τα συστήματα IT μεγάλης κλίμακας σύντομα θα έχουν ε, ένα νέο οργανισμό. Στο Ταλίνο όλα πηγαίνουν ρολόι σε αυτό το τομέα και περιμένουμε να κάνουμε τα εγγένεια του οργανισμού στα τέλη Μαρτίου στο Ταλίν. Τέλος, αυτή την τόσο σύντομη και πυκνή βεβαίως παρουσίαση λέγοντας ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική τη Ένωση για την εμπορία ανθρώπων περιμένουμε ότι θα τεθεί στο δεύτερο τρίμηνο τη χρονιά και θα είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτική με σκοπό την πρόληψη τη εμπορία ανθρώπων αλλά και την δίωξη όσων κάνουν τέτοια εγκλήματα και η προσοχή των θυμάτων και γνωρίζετε είναι κάτι που σα απασχολεί και σα βρίσκει ευαίσθητος. Λοιπόν, ε, πολύ πυκνό το πρόγραμμα εργασία μα. και όπως είπα στην αρχή Προσβλέπω ειλικρινά στη συνεργασία μαζί σας για όλα αυτά τα ζητήματα κατά το επόμενο διάστημα. Με αυτά τα λόγια, Πρόεδρε, ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Πιο σημαντικό βέβαια είναι να ακούσω τις ερωτήσεις για να έχουμε ένα ουσιαστικό διάλογο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας τους επόμενους μήνες. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τον κύκλο ερωτήσεων-απαντήσεων. Να ξεκινήσουμε τους συντονιστές. Each group then first round of answers and then... Μετά θα απαντήσει η Επίτροπος και μετά έχουμε το δεύτερο γύρο. Κλείνω τώρα τον κατάλογο, ούτως ώστε να προλάβουμε. Όπως έκανα και το πρωί ακριβώς. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι προβλέπουμε για αυτό το σημείο με την Επίτροπο, 50 λεπτά. Άντε το πολύ μια ώρα. Κάντε ό,τι μπορείτε για να μην να καθυστερήσουν τα επόμενα σημεία. Γιατί έχουμε τουλάχιστον άλλα 10 σημεία για την απαλλαγή, συν κάποια άλλα που πρέπει να διεκπαιρέωσουμε το απόγευμα. Και ξεκινάμε με ποιον άλλον, το Σάιμον Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Επ' θα ήθελα να σας ευχηθώ Καλή χρονιά. Ε, Ιανουάριος είναι ακόμα, μπορούμε να το πούμε νομίζω, να το λέμε μερικές μέρες. Ε, στο ΕΛΚ εμείς ετοιμιστήκαμε για αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής και ένα μείζον θέμα που έθεσαν τα μέλη μας είναι η τάση που βλέπουμε σχάτως για μια διακυβερνητικότητα ε, εις βάρος της μεθόδου, για να το πω έτσι. Το λέω καταρχήν, όχι γιατί μόνο πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, αλλά πιστεύουμε ότι και για σας είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να προτάξουμε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό για μας. Πρακτικά παραδείγματα που βλέπουμε αυτή την παρέκκληση θα έλεγα, είναι όχι μόνο η δημοσιονομική διάσταση, αλλά και ο χώρο έγκεν, όπου οι αντιδράσει δεν είναι ενθαρρυντικέ και σήμερα το πρωί μάλιστα συζητούσαμε το καθεστώ θεωρήσεων και τις αλλαγέ. Ε, καθώς και την ρήτρα διασφαλίσεων ή και το μηχανισμό αναστολής. Ακόμα και εκεί φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουμε ένα κοινό καθεστώ θεωρήσεων. Και αν μία ή περισσότερε χώρες μπουν σε ένα κατάλογο από μία τρίτη χώρα, μένουν μόνες τους στο κρύο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κοινωνική υποστήριξη. Η στάση είναι διακυβερνητική. Μιλάμε για, επίσης για αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου. Μιλάμε για ένα κοινό σύστημα ασύλου ευρωπαϊκό. Όταν όμως μια χώρα έχει δυσκολίες, μένει μόνη της. Είδα ένα άρθρο που γράψατε στην εφημερίδα μας Άρα σας απασχολεί, το ξέρω. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή η Κομισιόν τώρα να δείξει ηγετική τάση, να ανασχέσει αυτή την τάση διακυβερνητικότητας και να επιβάλλει την κοινοτική μέθοδο. Για την αλληλεγγύη. Ο Υπουργό ε, Δικαιοσύνης της Δανίας σήμερα το πρωί μας είπε ότι αύριο θα παρουσιάσει το θέμα, θα βάλει μάλλον το θέμα της αλληλεγγύης στην ατζέντα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Διερωτώμε αν η Κομισιόν έχει να κάνει ή θα κάνει συγκεκριμένη πρόταση, ούτω ώστε να πάρει σάρκα και οστά αυτή η, θα κανει συγκεκριμενη προταση ουτω ωστε να παρει σαρκα και ωστα αυτη η αλληλεγγύη. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, είχαμε την ανακοίνωσή σας για την αλληλεγγύη και σήμερα το πρωί ε, ο Διευθυντής της ΕΑΖΟ μα είπε ότι επίσης ε, συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε να, σύρε, να σηκώσετε αυτό το πέπλο μυστηρίου που υπάρχει σε αυτό, γύρω από αυτό το μηχανισμό αλληλεγγύης και να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Ε, σταματώ εδώ για να μην ξεπεράσω και το χρόνο μου. Δύο λεφτά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει ο καθένας σας. Βοηθήστε μας σας παρακαλώ, ούτω ώστε να επωφεληθούμε και από το δεύτερο γύρο ερώτα αποκρίσεων. Αν ο καθένας δείξει αυτοσυγκράτηση, όλοι θα μπορέσετε να μιλήσετε. Από εσά εξαρτάται, από τον καθένα δηλαδή από εσά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη γρήγορη επισκόπηση που μας κάνατε. Καλύψατε τόσο, τόσα πολλά θέματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ερωτήσεις. Καταρχάς, και εμείς έχουμε ανησυχίες για αυτές τις ε, διακυβερνητικές αποφάσεις και περιμένουμε να ακούσουμε την απάντησή σας στην ερώτηση Μπουσουτήλ. Πώς θα διαφυλάξετε την κοινωτική μέθοδο. Κάποια από τα θέματα που αναφέρετε είναι η συμφωνία με τους Αμερικανούς για το PNR. Είπατε ότι υπάρχει σοβαρή βελτίωση. Εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας ακούω ακόμα ανησυχίες για το αντίθετο. Υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια λιγμών στο μέλλον, ούτω ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη συμφωνία PNR. Πώ έχουν τα πράγματα σήμερα σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία. Για τη συνάντηση με τον Καναδά. Θα γίνει σήμερα το απόγευμα, είπατε. Δεν μπορείτε να προδικάσετε την συνάντηση που θα λάβει χώρα μετά αλλά θα ήθελα να μας πείτε περισσότερο για τα θέματα που θα καλύψετε. Υπάρχει σε εκκρεμή κατάσταση αυτή η υποχρέωση για τις θεωρήσεις. Ε, θα συζητηθεί αυτό σήμερα το απόγευμα. Μπορείτε να μας πείτε. Τρίτο ερώτημα. Ξεκινάτε το διάλογο για τις θεωρήσεις με την κυβέρνηση του Κόσοβο. Πήγατε πρόσφατα στη χώρα αυτή. Τι εντυπώσεις έχετε, πώς εξέλισω τα πράγματα στο Κόσοβο. Ευχαριστώ κυρία Γκούνς. Ε, καλωσορίζω τον κύριο Ντεκαπιτάνη. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ. από τους φιλελεύθερους κυρία Βέμπερ. Βέβαια. Ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, κάθε φορά που σας λέμε να έρθετε, ερχόσαστε. Το εκτιμούμε αυτό. Εκτιμούμε ότι είσαστε διαθέσιμοι. Θέλετε να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα. Και πριν και τώρα, χειρίζεστε ευαίσθητα θέματα. Ευαίσθητα. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει κατά ανάγκη σύμπτωση απόψεων Κοινοβουλίου, Κομισιών και Συμβουλίου. Ξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα για, θέματα, για τα θέματα του πακέτου μετανάστευσης και ασύλου. Αλλά δεν έχω την ίδια εμπιστοσύνη ότι θα περάσουμε όλα τα δικά μας θέματα. Είμαστε όμως να συμβαστούμε επικοδομητικά, αν τα καταφέρουμε. Και για την ενιαία άδεια βέβαια, αν μπορέσουμε. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο σημείο συνεργασίας. Βλέποντας τα θέματα που αναφέρατε και το πόσο σημαντικά είναι, μου έρχεται η εξής ερώτηση στο μυαλό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την ε, εντύπωση ότι εκπροσωπούμε διαφορετικούς ανθρώπους. Αλλά κανονικά και εσεί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εκπροσωπούμε του Ευρωπαίου πολίτε. Παραδείγματο χάρη για την οδηγία για τη φύλαξη στοιχείων. Είμαι σίγουρη ότι δεν τη θέλει το Συμβούλιο. Και όμω, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών ζητούν αλλαγή, πραγματική αλλαγή. αλλά φοβούνται μήπως η αλλαγή αυτή ε, πλήξει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Κάτω τους φιλελεύθερους θα μπορούσατε να είσαστε εκπρόσωπος που να εκφράζει τις απόψεις για την ιδεώδη συνεργασία που θα έπρεπε να έχουμε το Συμβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο θα έπρεπε κανονικά να σέβεται το Κοινοβούλιο και να σέβεται το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν και πιο δύσκολα θέματα και για το Κοινοβούλιο. Φυσικά είναι το PNR μεταξύ αυτών. Κυρίως συμφωνία PNR με τις ΗΠΑ. Δεν θα είναι εύκολο αυτό το θέμα για να κλείσει. Γενικά όμως έχει χωρίς αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Κυρία Σαρτζεντίνη από τους πράσινους. Ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο είναι η στρατηγική και την εσωτερική ασφάλεια. Έχουμε ένα σχέδιο κειμένου. Υπάρχει ένα σχέδιο που έχει ετοιμάσει ένα συνάδελφος. Ε, πίτροπε, αυτή η στρατηγική με ανησυχεί ότι οι στόχοι δεν είναι σαφείς, οι πληροφορίες ε, πάνω στις οποίες ε, βασίζεται δεν είναι ξεκάθαρες. Πρόσφατα ε, έχουμε δει κάποια ανάλυση από τη Europol που λέει ότι η απειλή είναι εξωτερική και είναι ισλαμικής φύσεως και προέλευσης. Όμως στην Νορβηγία είδατε τι έγινε. Είδατε τους φόνους που έγιναν από ακροδεξιού στη Γερμανία. Τον ακούμε ότι η στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια α, βασίζεται σε κάποιες απειλές που κανένας δεν ξέρει ποιες είναι και πώς αναλύονται κτλ. Αυτό μας ανησυχεί. Δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος αυτών των οργανώσεων που σας δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Ακόμα χειρότερο, είναι ότι αυτή η στρατηγική βασικά είναι στρατηγική καταστολής. Δεν θέτει θέματα δικαστικά, θεμελιωδών δικαιωμάτων, δικαστικής συνεργασίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη τα λύνουμε δήθεν με την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τη λέμε συνέχεια, την έχουμε καραμέλα και την πιπιλάμε, αλλά δεν λειτουργεί τόσο καλά. Υποτίθεται ότι έτσι εξασφαλίζουμε τους πολίτες μας από τις αυθαιρεσίε των κυβερνήσεων. Το πρόβλημα της στρατηγική είναι ότι εστιάζουμε συνέχεια στα εξωτερικά σύνορα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι βασικό εργαλείο για την ασφαλειά μας. Εσείς είσαστε Επίτροπος και Ασύλου και Μετανάστευσης και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα των συνόρων και της προστασίας τους. Ε, γίνεται μια συζήτηση για τα εσωτερικά σύνορα και το Σέγγεν και όμως θεωρούμε ότι με το να δίνουμε έμφαση στα εξωτερικά σύνορα και στη μετανάστευση κρατάμε έξω την απειλή και τον κίνδυνο. Είναι ατελής αυτή η στρατηγική. Βασίζεται σε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Τελευταίο σχόλιο, Πρόεδρε. έκθεση που έχει ετοιμαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτές τις ε, έκτακτες πτήσεις και κρατήσεις από την CIA ε, έγιναν ανταλλαγή μεταξύ Κομισιών και Κατών μελών. Καλό θα ήταν να δούμε αυτή την αλληλογραφία. Θέλω παρακαλώ να γίνει μια σωστή έρευνα και, μια, και να προκύψει μια καλή έκθεση για αυτές τις πτήσεις της CIA. Ο κ. Κύρκοφ. Κύρκοπ. Σύντομα. Μ' αρέσει η βασική ιδέα του προγραμματός σας, η ουσία του προγραμματός σας. Με ικανοποιεί εμπολής. Θέλω κάποιες διαβεβαιώσεις από την Κομισιόν ότι σε κάποιους δύσκολους τομείς όπου προσπαθείτε να εναρμονίσετε το σύστημα για σε κάποιους τομείς, με κάποια νομοθετήματα. Αν κρατήσουμε την ορμή που ε- υπάρχει ήδη στην ε, συνεργασία, γιατί δεν αρκεί αυτό για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι η πρώτη φάση. Εκεί είναι επιθυμητή για να πετύχουμε κάτι. Θα υπάρξει λοιπόν, θα κρατήσετε την πίεση για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία για σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά είναι η κυβερνοασφάλεια. Αναφέρεται στο πρόγραμμα ως νέα πρόκληση. Δεν είναι και τόσο νέα πια. Την αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό. Και η ζημιά που έχει γίνει ε, λόγω της παραβίασης της ασφα... κυβερνοασφάλειας είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, αλλά είναι ουσιαστική για και πλήττει ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τα άτομα και τις εταιρείε, αλλά και τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα η Κομισιόν να δείξει αποφασιστικότητα εδώ. Χρειαζόμαστε καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Ε, θα πρέπει να δουλέψετε και σε συνεργασία με τους Αμερικανούς διατλαντικά και να συνεργαστείτε και με άλλες χώρες όπου βλέπετε ότι υπάρχουν κρούσματα και όπου το θέμα αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Κάνω λοιπόν μία έκκληση. Τέλος. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία είναι κάτι που αναφέρεται. Άλλη έκκληση. Μπορούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία όπου μπορούμε, σας παρακαλώ και στην Κομισιόν, αλλά και αλλού. Γιατί μας βαραίνει πάρα πολύ η γραφειοκρατία, οι νόμοι, οι κανόνες. Νομίζω η Ευρώπη θα επωφελούνταν αν υπήρχε λιγότερη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Μποργέζιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι επίκαιρη. Συνέβησαν δύο πράγματα στη χώρα μου που δείχνουν κάποια πράγματα που στο παρελθόν ε, τα είχα επισημάνει και με ρωτήσεις εγώ προσωπικά. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν από αυτά που είπε δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά, γι' αυτό θα τα θέσω. Κατά τη διάρκεια της ε, διαμαρτυρίας των οδηγών στην Ιταλία ε, προέκυψε ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός από εταιρείε ξένες μεταφορικές κτλ. Που κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά με συνθήκες τελείως διαφορετικές. Σε επίπεδο κοινωνικό, ασφαλιστικό κτλ. Και με διαφορετικούς κανόνες από αυτούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σοβαρό. Γιατί υπάρχει όχι μόνο αθέμητο ανταγωνισμός, αλλά δημιουργούνται και κίνδυνοι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το ίδιο θα έλεγα και με τα πρόσφατα γεγονότα για το κρουαζιερόπλιο. Υπάρχουν εργαζόμενοι που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαβατήρια που εκδίδονται από τη Βουλγαρία και Ρουμανία σε ε, πολίτες τρίτων χωρών, όμορων τρίτων χωρών. Δεν θα έπρεπε να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη αυστηρότητα αυτά τα γεγονότα, γιατί δημιουργούνται κίνδυνοι, σοβαρότατα προβλήματα και, και βλάπτουν και τους Ευρωπαίους ε, εργαζόμενους. Χθες, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατήγγειλε Κάτι που συνέβη με την Ιταλική δικαιοσύνη, γιατί υπήρξε μια απόφαση για κάποιον ο οποίο μάλιστα ε, ήταν, είναι βουλευτής, μια κυρία, θεωρήθηκε ότι είναι, είπε πράγματα αντισημητικά και καταγγέλλεται ως προπαγάνδα αντισημιτική αυτό που είπε η κυρία αυτή. Κυρία Επίτροπε, γνωρίζετε αυτά τα πράγματα. Αντί να καταγγείλετε την συγγραφέα του Φιλαδίου, στην πραγματικότητα ε, καταγγέλλεται τον διευθυντή της εφημερίδας. Αυτή η καταγγελία έγινε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τύρι γίνει Χθίος Ε, για αυτό το θέμα της ε, αντισημιτικής προπαγάνδας που φοράει το μανδύα της σάτυρας. Λοιπόν, η κυρία Μάρσμου θα απαντήσει και μετά μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο που θα πρέπει να είναι πιο σύντομος από τον πρώτο. Ευχαριστώ για τα ερωτήματά σα. Όντω, κύριε Μποσότελ και εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η τάση της, που κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Το είδαμε τι συμβαίνει και με τη νέα οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε. Μάλλον θα χρειαστούμε πολύ περισσότερη Ευρώπη για να βγούμε από την κρίση. Αλλά δυστυχώ υπάρχει μια τάση να πάμε προ την άλλη κατεύθυνση. Τα κράτη-μέλη λοιπόν και οι εκλεγμένοι ηγέτε του θα πρέπει να συμφωνήσουν ε, σε κάποια πράγματα. Κάποια ήδη έχουν συμφωνηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει όντω καλύτερη υποπτία, καλύτερο έλεγχο οικονομικό. Είναι επικίνδυνη η τάση αυτή όμω που αναπτύσσεται και γι' αυτό η κοινότητα και τα θεσμικά του όργανα και η ε, Κομισιόν και το Κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία. Βλέπουμε πώ συζητώνται οι προτάσει που αφορούν τη Σέγγεν. Η Σέγγεν είναι ένα το μεγαλύτερο επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιο μίλησε για τους πολίτες. Αυτό πρέπει να το, ε, να το υποστηρίξουμε, να δούμε τι καλό έχει κάνει και να φροντίσουμε να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Να μην καταχρώμεθα τις ε, συνθήκες του Σέγγεν μόνο για εσωτερικού λόγους ή για προπαγάνδα. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε στενά. Για την αλληλεγγύη. Ξέρετε ποιε είναι οι απόψει μου. Η Κομισιόν παρουσίασε μια ανακοίνωση για την αλληλεγγύη λίγο πριν τα Χριστούγεννα και αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο θα συζητήσουμε αύριο το πρωί στην, στο άτυπο Συμβούλιο Τζάι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η ιδέα αυτή και την έχει αναλάβει σοβαρά η ε, Δανική Προεδρία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διατρεμιστικότητα γι' αυτό και ελπίζω ότι θα είναι και η φιλοδοξία τη Δανέζικη Προεδρία, αυτό το είπε και ο Υπουργό σήμερα, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτέ τι συζητήσει. Να μην μιλούμε μόνο θεωρητικά για την αλληλεγγύη, αλλά να έχουμε και κάποιε πράξει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξουμε την αλληλεγγύη μα. Τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι πολύ ενεργά όταν προσπαθούν να βοηθήσουν ας πούμε, την Ελλάδα. Ε, συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές για το σχέδιο δράσης, για το σύστημα ασύλου. Ε, βοηθούν με υπερογνωμοσύνη, με χρήματα, με κονδύλια. Θέλουμε να τα ενθαρρύνουμε να κάνουν κι άλλα. Θέλουμε να τα ενθαρρύνουμε να υποστηρίξουν την ΕΑΣΟ δίνοντας και την εμπειρογνωμοσύνη τους όταν αυτό χρειάζεται. Και επίσης θέλουμε να προτείνουμε ένα είδος πιο, πιο μόνιμου μηχανισμού ανακατανομής των κονδυλίων ε, έχουμε ευχαριστήσει βεβαίως τα κράτη-μέλη που ενεργά βοηθούν. Ξέρετε όμω ότι το έχω ξαναπεί. Δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Πρέπει να βάλουμε κονδύλια στο τραπέζι για να ενισχύσουμε τα κρατημέλη να κάνουν το ίδιο. Και μακροπρόθεσμα. Στι μακροπρόθεσμε προτάσει μα βάζουμε ε, λεφτά ώστε να μπορούν και τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν τη δική του επίδειξη αλληλεγγύη όχι μόνο όταν υπάρχουν οξύε κρίσεις, αλλά και σε καιρού ειρηνή ας πούμε, και σε πιο ε, φυσιολογικέ συνθήκε. Ο πρόεδρο θα είναι εκεί στη συζήτηση αύριο και φαντάζομαι ότι θα λάβουμε και την άποψη του Κοινοβουλίου προ αυτό, αυτό και βεβαίω μετά μπορεί να σα πει τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο. Η Προεδρία επίση ε, θα καταλήξει σε συμπεράσματα, όχι αύριο βεβαίω γιατί το Συμβούλιο είναι άτυπο, αλλά σε ένα επίσημο Συμβούλιο. Τώρα, κυρία Γκιόντ, για το PNR με τη ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση στο πεδίο εφαρμογή, στους ορισμούς, στην προστασία των δεδομένων, στις δυνατότητες που υπάρχουν για τους πολίτες να προσφύγουν. Το πεδίο τώρα χειρισμών που έχουμε είναι περιορισμένο. Δεν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε παραπάνω. Ε, αυτή είναι η συμφωνία και την έχει υποστηρίξει το Συμβούλιο. Αυτό την ξεκίνησε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν κάτι. Αυτό υπάρχει τώρα πλέον ως συμφωνία. Για τον Καναδά Νομίζω ότι είναι στην ε, ημερήσια διάταξή σας να σας ενημερώσει ε, αργότερα ένας προσεκλημένος για το πού έχουμε πάει με την συμφωνία με τον Καναδά, πού υπάρχουν δυσκολίες ακόμη. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα με τις θεωρήσεις ε, από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Εξακολουθεί να τρέχει ο διάλογος με τους Καναδούς. Δεν έχουμε ακόμα ότι δεν πηγαίνει γρήγορα, αλλά αυτή είναι η απόφαση. Γίνονται κάποιοι διάλογοι. Έχω συναντηθεί εγώ με τον Υπουργό αρκετέ φορέ για να το θέσω το θέμα αυτό. Για το κοσυφοπαίδιο τώρα, όταν ξεκινήσαμε το διάλογο, ε, το κάναμε με μεγάλη χαρά και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι το Κοσμοπέδιο δεν είναι πλέον απομονωμένο στα Δυτικά Βαλτάνια. Έχουν και αυτοί μια ευρωπαϊκή προοπτική και θα, το, θα, το, θα δούμε την περίπτωσή τους όπως κάναμε και με τους υπόλοιπους. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο Συμβούλιο, θα το συζητήσουμε, θα βρούμε έναν οδικό χάρτη όπως έχουμε κάνει με τις υπόλοιπες χώρες και με τη βάση, επί, επί της βάσης Βεβαίω ο οδικό χάρτη υπάρχει, αλλά θέλουμε να υπάρξει και μια τελευταία συμβολή από το ε, Κωσυφοπαίδιο και από το EULEX και από, τα από του υπόλοιπου ε, ε, εμπλεκόμενου φορέ. Ελπίζουμε λοιπόν επί τη βάση αυτή να μπορέσουμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσει αρχέ τη Άνοιξη. Βεβαίω ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποια σχέδια δράση για τη διαφθορά, την αντιμετώπιση τη κτλ. Βεβαίω, από εκεί και πέρα εξαρτάται από του ίδιου πόσο θα κρατήσει αυτή η προσπάθεια. Θα το κάνουμε όμω με ενδελεχή τρόπο όπω το έχουμε κάνει για όλου του υπόλοιπου έτσι ώστε να υπάρχουν και αυτοί, να έχουν και αυτοί μάλλον μια ευρωπαϊκή προοπτική και να μην αφήσουμε το ε, πεδίο απ' έξω. Κυρία Βέμπερ, ναι, όλοι δουλεύουμε για του πολίτε. Δεν νομίζω ότι βεβαίω οι πολίτε τη Ευρώπη έχουν την ίδια άποψη για τα πάντα και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Αλλά ο στόχο μα είναι αυτό, να ακούμε του πολίτε μα. Τώρα, για την ε, διατήρηση των δεδομένων, έχουμε την, ε, τα όσα προβλέπει το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη, λέει ότι τα, η διατήρηση δεδομένων και η δυνατότητα της αστυνομίας να βρει πώς ε, δρούν οι ε, λαθρέμποροι ναρκωτικών κτλ. είναι πάρα πολύ χρήσιμο ε, ως εργαλείο, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με την οδηγία αυτή που έχει να κάνει, έχουν να κάνουν με το πεδίο εφαρμογής ποιο μπορεί να, να χρησιμοποιήσει αυτή την οδηγία, χρονικά όρια κτλ. Ε, και αυτό προσπαθούμε εμείς να προτείνουμε στο Συμβούλιο να αλλάξει. Ελπίζω η συνεργασία μας να είναι καλή με εσάς, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κυρία Σαρτζεντίνη, το θέμα είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον ε, τομέα της ασφάλειας. Έχουμε δει ότι είναι το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα, το θέμα των συνόρων μας και διάφορε καταστροφέ. Ευρεία τη ενία, για να το πω έτσι. Το οργανωμένο έγκλημα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ ακριβεί στην, στην ανακοίνωσή μα, ώστε να θέσουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, η ε, αυξημένη αντιμετώπιση τη ε, διαφορά, κατάσχεση των, των κλοπημαίων. Ε, συμφωνώ μαζί σα βεβαίω ότι πολύ διστακτικά θα σας πω ότι έχουμε αποφύγει τις απειλές ε, και γι' αυτό ε, έχουμε ξεκινήσει και, το, ε, και, την, και την κίνηση αυτή κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Ξέρετε τι έγινε στην Ουτόγια, δεν θέλουμε να δούμε άλλα τέτοια συμβάντα όπως στην Νορβηγία. προσπαθούμε να ε, αποφύγουμε, να αντιμετωπίσουμε τη βία από νέων ή άλλων ατόμων που βρίσκονται σε πολύ ριζοσπαστικού κύκλου. Προσπαθούμε να του βγάλουμε από αυτόν τον κύκλο και να χρησιμοποιήσουμε την ε, εμπειρία που υπάρχει ώστε να αποφύγουμε ή να, προ, να προλάβουμε τον ε, ακραίο, την ακραία ριζοσπαστικοποίηση. θέλουμε λοιπόν να ενώσουμε τι δυνάμει μα, να ενώσουμε την γνώση που έχουμε. Κάποιε χώρε έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, κάποιε άλλε λιγότερο. Πρέπει λοιπόν να μοιραστούμε τι εμπειρίε μα, να κάνουμε κάποιε κοινέ προσπάθειε, να έχουμε πολύ περισσότερε προφορίε για το πεδίο ε, αυτού του εγκλήματο και πώ μπορούμε να προστατευτούμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η ε, προσπάθεια για το εγκλήμα, για τα σύνορα το να διαχειριστεί κανεί τα σύνορα είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Βεβαίω, ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε στο να, πιο ε, ευρία, να έχουν πιο ευρεία προσέγγιση, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην ε, που πρέπει να μην μπορούν να ε, εισέλθουν. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά εργαλεία για να ελέγξουμε τα σύνορα, να τα κλείσουμε σε εισαγωγικά. Βεβαίω πρέπει να αφήσουμε ελεύθερα τα σύνορα για του καλόπιστου επιβάτε, ταξιδιώτε, αλλά πρέπει να μην ανοίξουμε πολλά παραθυράκια ώστε να μπορούν οι άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματο να εισέλθουν. Επίση, υπάρχουν και άλλα σημεία που είναι μεγάλε προκλήσει, αλλά η στρατηγική για την ασφάλεια είναι να ερχόμαστε πάντα σε εσά, να ε, μπλέκεστε ε, ενεργά σε όλη τη διαδικασία, να σα αναφέρουμε πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν και τα θέματα ασύλου και μετανάστευση. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν παράλληλα. Κύριε Κέρκοπ, να πω ότι συνεργαζόμαστε με, τους, με τη ΣΥΠΑ, έχουμε τέσσερις ομάδες εργασίας για το κυβερνοέγκλημα και έγινε, υπευλήθη η πρώτη ετήσια έκθεση, θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας μαζί τους για να δούμε αν μπορούμε κοινά, κάποιες κοινέ ε, δοκιμές. Βεβαίω πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την παιδική προγραφία στο διαδίκτυο και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. και ο κύριος Ναπολετάνο έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει ενεργά στην ομάδα αυτή. Θα δούμε λοιπόν πώ μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να τον καλύτερα για τον κύριο Ποργιέζη, Ε, δεν γνώριζα αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, την ζωγραφιά αυτή που αναφέρατε, το φυλάδιο. Βεβαίω η Κομισιόν πάντα προσπαθεί να καταγράφει όλε τι περιπτώσει ε, ε ξενοφοβία, ομοφοβία, ε, δηλώσει αντισημιτισμού κτλ. Ε, το γεγονό ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το γνώριζα δεν σημαίνει ότι δεν το έχει καταγράψει η Κομισιόν. Αυτά και σα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ είναι περίπου 4 παρα 5. Που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα 12 που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο μόνος τρόπος για να πάρουν το λόγο και να έχουμε και απαντήσεις από την Επίτροπο είναι ο καθένας να μιλήσει μόνο, μέχρι, ε, να μιλήσει μόνο 1,5 λεπτό γιατί αλλιώς ή δεν θα μιλήσετε ή δεν θα πάρετε απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την πολύ ευσύνοπτη και πυκνή σας παρουσίαση και να σας πω ότι σίγουρα θα σας υποστηρίξουμε. Συγκεκριμένο ερώτημα. Ένα νομικό εργαλείο για την καλή διαχείριση της ε, μετανάστευσης είναι η πολιτική θεωρήσεων. Ένα εργαλείο, έτσι. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την τροποποίηση του κανονισμού 539 2001. Δύο λοιπόν ουσιαστικά ζητήματα τίθεται σε αυτή την τροποποίηση. Η ρήτρα υποχρέωση σε θεωρήσει μπορούμε να επιβάλλουμε στι δεύτερε χώρε έναντι καταχρήσεων, παράρτημα 1 και 2. Και το πλέον σημαντικό και έχει μεγάλη πολιτική διάσταση και για το οποίο θα ήθελα να ασχοληθεί περισσότερο είναι η αυτόματη αμοιβαιότητα. Τι σημαίνει με απλά λόγια. Αν μια τρίτη χώρα απαιτήσει, ε, επαναφέρει, επιβάλλει την υποχρέωση θεωρήσεων έναντι ενός κράτους μέλους, τότε και 27 θα πρέπει να αντιδράσουν ε, με τη μορφή του κατεπίκοντος. Και αυτόματα, ε, το υπογραμμίζω, αυτόματα και σε αλληλεγγύη ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και θα λαμβάνει η Επιτροπή αυτή την αυτόματη διαδικασία. Είναι μια μακρά συζήτηση αυτή που γίνεται λίγο τέτοιους μήνες και έχει λάβει και μεγάλη ε, δημοσιότητα και παρακαλώ το σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το πρόβλημα ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ε, φεύγουν ή αποστρέφουν το πρόσωπό τους από την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε καλύτερη κληρονομιά προς τον παρόν, την καταργούμε από μόνοι μας. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα με τη Σέγγεν. Τι γίνεται με την Ολλανδία όταν ας πούμε ε, γίνονται, βγαίνουν φωτογραφίες από ε, οχήματα τα οποία περνούν. Τι γίνεται με αυτές τις φωτογραφίες. Δεν μου έχει απαντήσει ποτέ κανεί. Η αλληλογγύη για τα κράτη-μέλη για τα εξωτερικά μα σύνορα επίση είναι σημαντική. Αλλά όλα τα κράτη-μέλη πάντα έχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολε καταστάσει να αντιμετωπίσουν. Εγώ έχω ε, πάει πολλές φορές σε τέτοια κράτη και δεν δίνεται πάντα η εντύπωση ότι έχουν τόση πολλή δουλειά που δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Ε. Τώρα, η συμφωνία PNR με τη ΣΥΠΑ μπορεί όντω να μπορούν να γίνουν βελτιώσει. Αλλά το ότι είναι καλή η, η συμφωνία αυτή σε σχέση με την παλαιότερη δεν σημαίνει ότι είναι και εξαιρετική. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν αυτέ οι βελτιώσει είναι περιφερειακά σημεία ή αν είναι κεντρικά σημεία. Και ένα τελευταίο θέμα για την προστασία των δεδομένων και την αποθήκευση των δεδομένων. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να αλλάξουν ε, κάποια πράγματα. Αυτό όμω δεν μπορεί να γίνει, να αποτελέσει για μα αντικίνητρο για να, μην, για να κάνουμε μόνο ελάχιστε αλλαγέ. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για πραγματικά ελάχιστε, ε, μικρά, πολύ μικρά ε, αδικήματα. Αν τώρα αυτή η οδηγία θέλει να μπει και στα πλαίσια της, ε, του της ανταγωνιστικότητας, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τίποτα με, τους, ε, με την προστασία των ε, δικαιωμάτων των πολιτών. Ο κύριος Κοέλιο. Ε, και εγώ να σας συγχαρώ για την πρώτη τοποθέτηση και για το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, η αξιολόγηση του συστήματος Schengen. Μια χρονική στιγμή όπου τα κράτη τη μελη ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να υπάρχει συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Κύριε Επίτροπε, έχετε την... εμένετε στην ίδια στάση που είχατε τη αρχή, Εμείς χειροκροτούμε την πρωτοβουλία σας και την νομική βάση του άρθρου 77. Ρωτώ κατά πόσον κρατάτε την ίδια γραμμή μετά την ιδρύση του Συμβουλίου. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά πρόβλημα με τη δεύτερη γενιά του συστήματο SIS. Η κυρία Επίτροπο μπορεί να μα επιβεβαιώσει ότι το 2013 θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα ή θα έχουμε καθυστερήσεις για την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρία Φάγιαν, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, Κύριε Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω και εγώ για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων, ιδίως η έναρξη του διαλόγου για το κοσφοπέδιο. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας εν προκειμένου, αλλά θέλω να ρωτήσω μια λεπτομέρεια για αυτό το θέμα. Ο δικός χάρτης για την Πρίστρια, δηλαδή Πότε νομίζετε ότι θα ελεγχθεί ο οδικό χάρτη και θα υποβληθεί στι αρχέ του κοσμοπεδίου. Άκουσα τα σχόλια από την Πρίστινα ότι αν είναι ο ίδιο οδικό χάρτη όπω και τι άλλε χώρε ειδικών Βαλκανίων, τότε θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί λόγω των γεγονότων στο βορρά τη χώρα. Οπότε η όλη διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει. Ποια είναι η γνώμη σα. Έπειτα, κοιτώντα τελευταία έκθεση τη Frontex, βλέπουμε ότι οι αιτήσει ασύλου από τις πέντε χώρες των Βαλκανίων που εξαιρούνται από θεωρήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Όμως στη δική σας χώρα το Δεκέμβρη, στη Σουηδία, είχαμε α, μεγάλη αύξηση των αιτήσεων ασύλου, ιδίως από Βοσνία Ερσεγοβίνη. Γενικά όμως είχαμε μείωση. Σε ό,τι αφορά την Σουηδία και ετούντες άσυλο από Βοσνία Ερσεγοβίνη, ρωτώ, θα λάβετε συγκεκριμένα μέτρα Έχετε κάποιες επαφέ με τη Σουηδική κυβέρνηση, τι προθίσετε να γίνει. Και όσον αφορά το διάλογο και την πολιτική θεωρήσεων, Ποια είναι η επόμενη χώρα στην γειτονιά τη Ένωση που θα μπει στο καθεστώ τη απελέγης θεωρήσεων. Τι προβλέπετε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται τα πράγματα να ειναι καπω κάπως στολά. Ευχαριστώ κύριο Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ την κύριε Επίτροπο για την παρουσίαση. Πέρυσι περίπου σας είχα πενθυμίσει ότι η Frontex για πρώτη φορά είχε μια στοχευμένη αποστολή με την ε, πολύ γνωστέ αποστολέ Rabbit στον Εύρο. Στόχο τη αποστολή αυτή ήταν ε, να αντιμετωπίσει τι μεγάλες ε, μεγάλους όγκους ροών παράνομων ταναστών που περνούν τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Είχαμε την ανακοίνωση της Επιτροπής της Frontex για τη μείωση των εισρωών το πρώτο δίμηνο, αν θυμάμαι καλά. Και λήφθη λοιπόν η απόφαση να παραμείνει η Frontex εκείνη την περιοχή με ένα project ονόματι Ποσειδώνας ώστε να υπάρξουν μόνιμες αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην περιοχή. Ένα χρόνο μετά, η εικόνα είναι η αντίθετη έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αριθμοί, πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι πριν την αποστολή Περίπου 320 άτομα ε, υπολογίζω ότι ε, μπαίνουν καθημερινά στο ευρωπαϊκό έδαφος, περνώντας τα συνορα ελλαδα Ελλάδας-Τουρκίας. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, δεν έχουμε επιτυχία σε αυτή την επιχείρηση που έκανε η Frontex. Για τέτοιου είδους λοιπόν παρεμβάσεις ο ρόλο τη Frontex είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για τη σημερινή παρουσία στην Επιτροπή μας και ζητώ από τον Προεδρό να μην υπολογίζει το χρόνο που θα μιλήσω. Ήθελα να θέσω κάτι της διαδικασία. Θα μπορούσε η Επίτροπος να επιστρέψει και το Φλεβάρι και το Μάρτι, γιατί με 1,5 λεπτό δεν προλαβαίνουμε να θέσουμε όλα τα ερωτήματα που μας απασχολούν. Παρακαλώ μην το καταλογίσετε στο χρόνο μου, πρόεδρε, αυτό που είπα. Τώρα ξεκινάω. Κυρία Μάλστρομ, σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δανό Υπουργό Δικαιοσύνη, όπως και τον εκτελεστικό διευθυντή τη ΕΑΣΟ στη Μάλτα. Και ρωτώ, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου τι εργαλεία θα του δώσει ώστε να λαμβάνει στοιχεία από τα κράτη-μέλη για τα κέντρα υποδοχή προσφύγων, ο οποίο μα είπε ότι δεν έχει καμία ευχαίρεια και καμία δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίε από τα κράτη-μέλη. Μα αν η ΆΣΟ δεν έχει πληροφορίε, τότε τι δουλειά θα κάνει. Μόνο κατάρτιση του προσωπικού που θα βρίσκεται στα κέντρα υποδοχή. Μα αυτό δεν ήταν ο σκοπό δημιουργία του ΕΑΣΟΝ. Μιλούμε για ένα κοινό σύστημα ασύλου. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορεί η ΕΑΣΟ να παίρνει πληροφορίε. Πόσα άτομα υπάρχουν στα κέντρα υποδοχή, πώ είναι το άσυλο, πώ είναι ο χρόνο αναμονή, διεκπαιρέωση τη αίτηση, ποιε είναι οι συνθήκε κράτηση κτλ. Και δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Το Γραφείο Ασύλου πρέπει να λαμβάνει πληροφορίε. Η Κομισιόν έχει δυνατότητα πρωτοβουλία εν προκειμένου να απαιτήσει να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίε ή η ΆΣΟ, διότι αυτό που μα είπαν το πρωί είναι ότι προσπαθούν μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων να αποσπάσουν πληροφορίε. Αυτό μου φαίνεται ασόβαρο. Ε, δεν θα μπορούσε αυτό να τεθεί και αύριο στο άτυπο συμβούλιο Τζάι. Δεν πρέπει και τα 27 και αύριο τα 28 κράτη-μέλη να δίνουν αυτές τις πληροφορίες στην ΕΑΣΟ. Ιδάλλως καταλήγουμε στα τυφλά, χωρίς πληροφορίες. Χωρίς πληροφορίες δεν υπάρχει καμία, ε, κανένα κοινό σύστημα. Και επειδή δεν έχω άλλο χρόνο να πω εντάχει, Πρόεδρο, το σχέδιο βοήθειας για την Ελλάδα. Σε τι συνίσταται. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, σε ό,τι αναφορά το περισμό του χρόνου, το θέτουμε για να μπορούν να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Ο πρώτος κανόνας που ισχύει στην Επιτροπή είναι ότι πάντοτε έχουμε βεβαρημένη ατζέντα. Δεύτερος κανόνας, όλα τα μέλη της Επιτροπής συνεχίζουν να πιέζουν, έχουμε και πιο πολλά ακόμη θέματα στη μεσαδιάταξη. Ε, άρα, πάντοτε ξεπερνούμε το χρονικό όριο που έχουμε και για να δώσουμε λοιπόν χρόνο σε όσο γίνεται πιο πολλούς αγορητές, γι' αυτό σας παρακαλώ να κρατάτε το όριο που σας δίνουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε πολύ πιο ευσύνοπτοι στην ε, τοποθέτησή σας, για να δώσουμε και χρόνο και στην Επίτροπο να απαντήσει. Ο κύριος Γιακολίνο. Θα είμαι συντομότατος. Ευχαριστώ την κυρία Μάλστρομ για την ε, διαθεσιμότητά της και την ε, μεγάλη ακρίβεια στην τοποθέτησή της. Η ερώτηση έχει ως εξής. Σε μια πρόσφατη ευκαιρία που είχαμε μια επαφή, συζητήσαμε τις συμφωνίες συνεργασίας με τις όμορες χώρες στα νότια της Ευρώπης για την ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών. Έχουμε κάποια καινούργια στοιχεία. Στην περίπτωση της Αιγύπτου την Τινησίας και Λιβύης έχουμε να κάνουμε με νέες έθραυστες δημοκρατίες. Αυτές οι συμφωνίες συνεργασίας δεν θα πρέπει κανονικά να συνομολογούνται εξ ονόματος Ένωσης και να μην έχουν διμερή χαρακτήρα. Όταν μιλούμε για αλληλεγγύη και για υπευθυνότητα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργούμε εύρωστους οργανισμούς. Ε, ό,τι έχουμε δημιουργήσει σήμερα δεν ε, μπορούν να μας επιτρέψουν να έχουμε μια ουσιαστική συνεργασία με αυτές τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε στην νότια πλευρά της Μεσογείου. Υπάρχουν ε, πολλές προθέσεις, αλλά παρά τα αυτά η Νότια Μεσόγειος ε, είναι ακόμη πηγή μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπότσκουρτ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Μιλήσαμε λιγάκι για την ακραδεξιά. Βλέπουμε τις πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ακραία δεξιά, η άκρα δεξιά, συγγνώμη, λειτουργεί ανενόχλητη και κάνει ό,τι θέλει ανενόχλητη. Την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Κοινοβουλίου ε, διαπιστώνει ότι ο αντισημιτισμός στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες ε, το φαινόμενο αυτό αυξάνεται. Τώρα, για την άκρα δεξιά, για τον αντισημιτισμό. Έχω υπόψη εδώ πέρα τις ε, δολοφονίες άκρας δεξιά στη Γερμανία. Θα κάνει η Κομισιόν κάποια έρευνα για αυτή την ε, τον πολλαπλασιασμό αυτού του φαινομένου στην Ευρώπη. Στο τέλος της Πολωνικής Προεδρίας έκανα το ίδιο ερώτημα στην Πολωνική Προεδρία. Αλλά μου είπε ουσιαστικά ότι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα η Πολωνική Προεδρία. Η Κομισιόν έχει την, την πρόθεση να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και κάτι πρέπει να γίνει. Δεύτερο σημείο, η οργανωμένη εγκληματικότητα. Μας είπατε ότι είσαστε έτοιμοι να κατασχέσετε προσόδους από οργανωμένη εγκληματικότητα από οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει ε, δυνατότητα για συνεργασία με όλες τις ε, αρχές, δηλαδή φο... Ε, φορολογικές αρχές, με το δασμολόγιο, όμω είναι υπεύθυνοι για το δασμολόγιο. Μερικές φορές είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε όλες τις κινήσεις των εγκληματιών αυτών. ευχαριστώ την Επίτροπο. Και αν γίνει και μάλιστα ε, θέλω να πω ότι έγινε προτεραιότητα η οργανωμένη εγκληματικότητα χάρη και σε εσά. Όταν προτείνετε το πακέτο για την ε, δίμευση ε, στη φάση εκπόνησής του λάβατε υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, η αξιολόγηση της απόφασης πλαίσιο της απόφασης πλαίσιο 8041, ε, πώς την αξιολογείτε, η κυρία Φλότχα. Κυρία Μάστρομ, σας ξέρουμε, συχνά κάνετε δηλώσεις ε, για θέματα όπως τον Κουαντάναμο κτλ. Ποια αξιολόγηση μου είπατε, δεν άκουσα το τέλος, κυρία Αλφάνο. Της απόφασης 2008 841. Τζάι. Είναι απόφαση πλαίσιο, λοιπόν. Μα λέτε απλώ το νούμερο. Τι απόφαση είναι αυτή, μπορείτε να μα θυμίσετε. Αφορά γενικά το πλαίσιο γύρω από το θέμα της οργανωμένης εγκληματικότητας. Έλα Τι γίνεται για αυτό το θέμα. Λοιπόν, Φλότρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κάνει μια δουλειά για αυτό το πρόγραμμα ε, έκτακτων πτήσεων της CIA. Οι ευρωβουλευτές θα χρειαστούν τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε κάνει σχετικά δηλώσεις, είστε γνωστοί γι' αυτό, χρήσιμες δηλώσεις. Θα ήθελα να εξασφαλίσω τη συνεργασία μαζί σας σε όλους τους τομείς για αυτό το θέμα σύντομα τώρα. Ε, με, Μεσόγειος, ε, πρόγραμμα για την κινητικότητα. Το πρόσωπο της Ευρώπης, ε, αυτό που είδαν όλοι οι άνθρωποι, είναι ότι διώχνουμε τους λαθρομετανάστες. Τι φιλοδοξία έχετε εσείς τι στάση θέλετε να κρατήσετε στις διαπραγματεύσεις με τις νέες δημοκρατικές χώρες, δηλαδή την Ισία ε, και τις υπόλοιπες χώρες της Νοτίου Μεσογείου, της Νότιας Όχθης Μεσογείου. Και τώρα η Επίτροπος Μάλστρομ για να απαντήσει συνολικά. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Δύο γενικές παρατηρήσεις. Κυρία Σαρτζεντίνη, δεν απάντησα προηγουμένως για την ε, CIA και η κυρία Φλότ επανέλαβε το ερώτημα. Ξέρετε πολύ καλά. Δούλεψα και στην ομάδα με το, του κ. Κουέγιο, Με ενδιαφέρει. Βασικά, ε, η αρχική πρωταρχική αρμοδιότητα είναι της ε, Αντιπροέδρου Ρέντινγκ. Αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα συνεργαστούμε και με τη Διεθνή Αμνηστία και το συζητήσαμε τις προάλλες με τη Διεθνή Αμνηστία. Ε, ούτως ή άλλως, ενδιαφέρουμε πολύ, θέλω να έρχομαι στην Επιτροπή και την επόμενη φορά μπορούμε να προβλέψουμε περισσότερο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις και λιγότερο για παρεμβάσεις. Είμαι στη διάθεσή σας. Κύριε, κύριε Στεμέρα, Μέρα, για την αμοιβαιότητα και τις θεωρήσει θεωρήσεις με τον Καναδά και τα λοιπά. Ξέρω πολύ καλά το πρόβλημα. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πνεύματος πάντα προσπαθούμε να βρούμε λύση πριν την αντιπαράθεση. Αυτή τη μέθοδο έχουμε χρησιμοποιήσει με τον Καναδά. Και πραγματικά είμαι απογοητευμένη με τους Καναδούς γιατί το πρόβλημα παραμένει εδώ και καιρό. Είναι απαράδεκτο ε, να επιβάλλονται τέτοιε υποχρεώσει θεωρήσεων για κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βρεθεί λύση. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε από πίσω όλο το Συμβούλιο. Δεν είναι μία απόφαση που μπορεί να πάρει μόνο η Κομισιόν. Κυρία Σίμπελ, για αυτά που συνέβησαν στην Ολλανδία και το Σέγγεν. Δύο φορέ γράψαμε σε Ολλανδικέ Αρχέ και ζητήσαμε πληροφορίε. Περιμένω ακόμα τις απαντήσεις των Ολλανδικών αρχών για το τι σκοπεύουν να κάνουν στα σύνορά του. Για την ελληνική, το ελληνικό θέμα έχουμε δώσει χρήμα και πόρους. Έχετε δίκιο. Στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ξοδεύονται σωστά τα χρήματα. Δεν δίνουμε απλώς χρήματα σε ελληνικές αρχές. Ε, τα δίνουμε για συγκεκριμένα έργα και project με την εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων αρχών. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν όπω πρέπει. Υπήρξε πρόβλημα και το έχουμε συζητήσει με τι ελληνικέ αρχέ. Δηλαδή, δεν υπήρξε δυνατότητα απορρόφηση όλων των κονδυλίων και εργαζόμαστε ακριβώ γι' αυτό. Δεν του δίνουμε απλώ επιταγή εν λευκό, του δίνουμε λεφτά για συγκεκριμένα project. Κύριε Κουέγιο, η Κομισιόν για προφανεί λόγου πρότεινε όλες οι αλλαγές στον κανονισμό του Σέγγεν να γίνουν με βάση το άρθρο 77 στην απόφαση. Δεν άλλαξαμε γνώμη, είναι σημαντικό αυτό γιατί αφορά και τα τρία θεσμικά όργανα, αλλά και γιατί αυτό που προτείνουμε στην αξιολόγηση, για την αξιολόγηση, είναι να μπορούμε να εντοπίσουμε εγκαίρως τα πιθανά προβλήματα και να συνεργαζόμαστε με το συγκεκριμένο κράτο μέλου για να βρούμε ένα σχέδιο δράση και τα εργαλεία, ούτω ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα, ούτω να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε το άρθρο 97. Δεν έχουμε, δεν έχουμε παραιτηθεί από αυτό. Ελπίζω και το Συμβούλιο να προχωρήσει. Γίνονται διάφορες συζητήσεις. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα της νομικής βάσης. Γίνονται παράλληλες συζητήσεις και ελπίζω παράλληλα να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τα του περιεχομένου, όχι μόνο το νομικό, ας πούμε, φορμαλιστικό θέμα. Επίσης έχουμε κάποια προβλήματα για τις θεωρήσεις. Ε, είχαμε επαφές με κάποια κράτη-μέλη, προσπαθήσαμε να τα υποστηρίξουμε. Και ελπίζουμε η δέσμευση που έχουμε αναλάβει όλοι να μας βοηθήσει ούτω ώστε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα του 2013. Δεν χρειάζεται προς το παρόν να αμφισβητήσουμε τη δέσμευση. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη όμω. Προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Κυρία Φατζάν, για το κοσφοπέδιο θα του δώσουμε τον ίδιο δικό χάρτη με του υπόλοιπου. Δεν είναι μόνο στα χέρια μου αυτό το θέμα, να αποφασίζω μόνη μου. Θα πρέπει να εμπλέξουμε και το Συμβούλιο. Δεν μπορώ να σα δώσω ημερομηνία. Ελπίζω να γίνει την άνοιξη αυτό. Φυσικά η διαχείριση των συνόρων είναι πολύ σημαντικό θέμα για τι θεωρήσει. Προφανώ δεν μπορούμε το. Είναι εκτό των Ουκάνεφ. Και βεβαίω θα λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε του Κόσοβο. Ε, ο διάλογος Πριστίνα Βελιγραδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρου ένα παράλληλο διάλογο. Και εκεί πρέπει να βρούμε λύση. Δηλαδή, η διαχείριση των συνόρων είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και γίνεται αυτό ο διάλογο. Ούτω ή άλλω, ε, συζητάμε ε, γενικά με όλε τι χώρε τη γειτονία αυτή. Ανατολική Ευρώπη και Νότια Ευρώπη. Κύριε Βανικολάου, Frontex. Το Δεκέμβριο το συζητήσαμε το θέμα αυτό. Ελπίζουμε να έχουμε μια νέα επιχείρηση Rabbit της Frontex, αλλά αυτό εξαρτάται από το αν τα διάφορα κράτη-μέλη θα μας δώσουν τους πόρους ε, για τη Frontex. Ελπίζω να δεχτούν. Ελπίζω λοιπόν να συνεργαστούμε περισσότερο με την Ελλάδα για το θέμα των συνόρων για να προχωρήσουμε το θέμα του Rabbit. Κυρία Ρομέρο Λόπες, σημαντικό το σημείο που θέσατε, θα το εξετάσω. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο μετανάστευσης όπου όλοι, όλα τα συμβούλια, τα ευρωπαϊκά, τα εθνικά συμβούλια μάλλον, δίνουν στατιστικές. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, θα το κρατήσουμε ψηλά στις προτεραιότητές μας και αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές θα τις κάνουμε. Γιατί δεν έχει νόημα χωρίς αυτές τις πληροφορίες. Κύριε Γιακολίνο, και εσείς και άλλοι ρωτήσατε για τους νότιους γειτονές μας οι εξελίξει δεν είναι ίδιε στι διάφορε χώρε. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά, είναι κατάλληλη στιγμή για να έρθουμε σε επαφή με του ανθρώπου αυτών των χωρών, των νότιων γειτόνων. Έχουμε μια εταιρική σχέση για την ασφάλεια και την κινητικότητα και εκεί θα καλύψουμε σε αυτό το διάλογο όλα τα θέματα. Τα θέματα ασύλου, ε, λαθρομετανάστευση, επιστροφής, επανεισδοχής, διευκόλυνση τη νόμιμη μετανάστευση. Ε, να δημιουργήσουμε ας πούμε, πιθανώς γραφεία σε αυτές τις χώρες για να τις βοηθήσουμε. Να διευκολύνουμε την κινητικότητα μέσω του διαλόγου για τις θεωρήσεις, αλλά επίσης και θέματα ασφάλειας. Να δούμε ας πούμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την αστυνομία στην Τινησία για να γίνει πιο δημοκρατική αυτή ας πούμε, η, η αστυνομία παρά να εξυπηρετεί μια δικτατορία. Μαρόκο, την Ισία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, αλλά μας ενδιαφέρουν και οι υπόλοιπε χώρες ανοίγουμε και σε αυτού. Ε, εξαρτάται πάντα από την κατάστασή τους. Πρέπει να έχουμε και έναν ομόλογο για να συζητήσουμε. Κοιτάξτε, ε, δεν μπορώ να σας πω πράγματα για τι συμφωνίε που κάνουν οι επιμέρους ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εκεί δεν υπάρχει τόση διαφάνεια. Κυρία Μπόσκουρ, δύσκολο το ερώτημά σα Δυστυχώ, ξέρουμε ότι ε, αυξάνονται τα κρούσματα επιθέσεων τη ακραδεξία. Ε, Κάναμε πολλέ συζητήσει στο Σώμα των Επιτρόπων για το θέμα αυτό και συζητήσαμε και με την ε, Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία προσπαθεί να χαρτογραφήσει την κατάσταση για να βρει παραδείγματα καταπολέμηση. Επίση, ε, προσπαθούμε να δούμε και παραδείγματα ε, αντίθετα από την ριζοσπαστικοποίηση. Ε, υπάρχει βεβαίως προπαγάνδα ε, υπέρ της άκρας δεξιάς, υπάρχει όμως και το αντίθετο Υπάρχουν και άλλες απόψεις στο ίντερνετ και προσπαθούμε να βρούμε, ας πούμε, φως εκεί. Είναι πολύ δύσκολο όμως να δημιουργήσουμε μια στρατηγική για την καταπολέμηση, ε, γιατί το θέμα είναι ποιος παίρνει τον ηγετικό ρόλο στις επιμέλους, επιμέρους χώρες, ε, ποιες κοινότητες, ποιες τοπικές αρχές. Ε. Βασικό είναι αυτές να μην συμφωνούν με τα θέσφατα της άκρας δεξιάς. Οι απαντήσεις μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Φλότρα, CIA. Απάντησα νομίζω. Ο διάλογος για την κινητικότητα αφορά και το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά φυσικά εδώ πρέπει να μας βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν δηλαδή. Ε, πρόεδρε, ελπίζω ότι κάλυψα όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον όπως είπα και στην κυρία ε, Λόπες Ρομέρο, Ρομέρο Λόπες μάλλον, ε, οποιαδήποτε στιγμή είμαι στη διαθεσία σας να επανέλθω. Εμείς αντίθετα σας ευχαριστούμε. Και όχι πρώτη φορά, για πρώτη φορά. Είχαμε προβλέψει μία ώρα και τώρα έχει περάσει μία ώρα και 20 λεπτά που το συζητάμε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει δύο ώρες. Αλλά ακόμα και τώρα Ακόμα και τότε, ακόμα και δύο ώρε να είχαμε προβλέψει, δεν θα φτάνε, θα υπήρχαν παράπονα, θα θέλατε περισσότερη ώρα, γιατί πραγματικά τα θέματα σα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σα ευχαριστώ για την καλή συνεργασία με την Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ που κάνετε ό,τι μπορείτε. Όχι μόνο για να είσαστε συχνά παρούσα και να κρατήσετε το διάλογο με τα μέλη μας, αλλά και να μας δίνετε πλήρης και ακριβή απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε να σας ξαναδούμε. Αν μου επιτρέπετε... Αν μου επιτρέπετε... Πάμε στο επόμενο σημείο χωρίς άλλες καθυστερήσεις γιατί έχουμε να συζητήσουμε καμιά δεκαριά απαλλαγές. Αλλά πρώτα θα δούμε τη στρατηγική για την ε, ιστορική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Ρίτα Μπορσελίνο έχει αναλάβει τη σχετική έκθεση, έγινε μια ε, συνάντηση την, τον προηγούμενο Οκτώβριο για την ευθύνη, για τον, ε, για το ρόλο της Europol, της Eurojust, Frontex και, τη, και έχουμε την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή όλων αυτών της Κομισιόν. Θα ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται, πώς έχει η κατάσταση και τι γίνεται με το σχέδιο κειμένου της έκθεσης της κυρίας Μπορσελίνο. Βεβαίω μετά θα κάνουμε και μια σύντομη συζήτηση. Ε, η αντιπρόεδρος Συνετφέλτ θα πάρει το... θα αναλάβει την Προεδρία για το επόμενο μισάωρο γιατί έχω μια υποχρέωση. Θα επανέλθω όμως μετά από αυτό το σημείο, θα επανέλθω. Okay. Um, thank you. We'll first give the floor. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μπορσελίνου. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί και αγαπητέ συνάδελφοι, θα σα παρουσιάσω σήμερα ένα σχέδιο έκθεση που είναι το αποτέλεσμα μια σειρά συνεδριάσεων που είχα με του κοιότε ηγητέ που του ευχαριστώ ευθύ εξ αρχή για τη συμβολή του και την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του ευρωπαϊκού οργανισμού. Μία διευκρίνηση στην έκθεση έπρεπε να λάβω υπόψη ε, και τους περιορισμούς ε, του ιστορικού κανονισμού για τον αριθμό των λέξεων που έπρεπε να χρησιμοποιήσω. Έτσι δεν μπόρεσα να εμβαθύνω περαιτέρω, ε, χρησιμοποιώντας όλες τις τροπολογίες που ευλήθην. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα θα κάνω μια στούμη παρουσίαση και θα παρουσιάσω τα πλέον σημαντικά στοιχεία της εκθέσης. Πρώτα απ' όλα, θέλω να επισημάνω ότι η ασφάλεια είναι ένα μείζον ζήτημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ρητά έχει δεσμευτεί για την εκπόνηση μιας ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την Ένωση. Η ασφάλεια όμως θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι αδιανόητο να ε, βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο. Η πραγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ουσιώδη συνιστόσα της πολιτικής ασφάλειας, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη ε, αυτό το σημαντικότατο άξονα στην προτινόμενη στρατηγική. Πολύ σημαντικός ο ρόλος προκειμένου των ευρωπαϊκών θεσμών στον καθορισμό και την υλοποίηση στρατηγικής, ιδίως με στα πλαίσια ε, μετά την θέσπιση της συνθήκης Λισαβόνας, ιδίως όταν αφορά πολιτικές μικτής αρμοδιότητας, θα πρέπει ε, βάσει της συνθήκης αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα κράτη-μέλη για την εσωτερική ασφάλεια. Άρα εκεί θα πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεπικουρήσει τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν εν προκειμένου να προβλεφθεί και ο κατάλληλο όλο του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την εκπόνηση προτεραιοτήτων στρατηγική αλλά και για την αξιολόγησή τη. Πρόκειται για ένα ρόλο που απορρέει από τον ρόλο του νομοθέτη που έχει αναλάβει πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα ασφάλειας. Επίσης, είναι ουσιώδε στοιχείο για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε επαρκή δημοκρατικό έλεγχο, κάτι που πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίπλα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει θεσμοποιημένη σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει ένα μόνιμο κύκλο που να συνδέεται με την ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό, που θα ολοκληρώνεται με μία ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου για το επίπεδο υλοποίηση στρατηγική εσωτερική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις, ε, τις απειλές δεν έχει γίνει μια σφαιρική ανάλυση προκοπέδου για την απειλή που αντιμετωπίζουμε με ομοιόμορφες παραμέτρους και με αξιόπιστα δεδομένα. Μόνο επί μια τέτοιας βάσης θα μπορούν οι συνομοθέτες να κινηθούν κατάλληλα. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες για να ορίσουμε καλύτερα τις παραμέτρους και κοινέ στατιστικές μεθόδους και την ανταλλαγή δεδομένων βάσει των οποίων κάνουμε την αξιολόγηση των απειλών κάνουν αξιολόγηση τα ευρωπαϊκά όργανα. Ιδάλλως θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε συνεχείς πιέσεις χωρίς να έχουμε μία κοινή στρατηγική. Σε ό,τι αφορά τις πέντε προτεραιότητες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρατηρείτε, διαβάζω την έκθεσή μου, ότι δεν ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για τον κάθε ε, επιμέρους στόχο διότι σε, ε, κάποιες πρωτοβουλίες είναι και άλλες ακόμη δεν έχουν υιοθετηθεί. Εγώ προσπαθώ να ακολουθήσω μια σφαιρική προσέγγιση στην εκθεσή μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξελικτικός ή τουλάχιστον και οι πέντε στόχοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ισότιμοι. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κλιματικότητας δεν μπορούν να θεωρούν ότι είναι το ίδιο πράγμα με τις θεομηνίες ή τις κατασπρόσεις που προκαλεί ο άνθρωπος, όπως επίσης η προστασία της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Βεβαίω είναι όλα ευαίσθητα ζητήματα. Το οργανωμένο έγκλημα, η καταπολέμηση τη δημοκρατία είναι δύο μέγιστε προτεραιότητε στρατηγική τρίτη ασφάλεια και οι στόχοι του θα πρέπει να αξιολογούνται όσο γίνεται πιο ορθά. Και αυτό μας το υπενθυμίσουν και τα ad ψηφίσματα που υιοθέτησε πρόσφατα το Κοινοβούλιο μα. Σε ό,τι αφορά την ριζοσπατικοποίηση, θεωρώ ότι μετά τα γεγονότα στην Νορβηγία και το δίκτυο των νεοναζί στη Γερμανία, ε, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα θρησκευτικό φανατισμό. Έχουμε να κάνουμε με ριζοσπαστικά κινήματα, πολύ βία, που έχουν ε, σαφή ιδεολογική χρειά και που αντίκειται στι αρχέ τη ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση, που βασίζεται όμω σε αυτέ τι αρχέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια των συνόρων στα πλαίσια της στρατηγικής για την ασφάλεια. Παρότι είμαστε γενικά υπέρ, θεωρούμε ότι η διαχείριση των συνόρων κινητικότητα των προσώπων δεν αποτελούν πρόβλημα ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα είναι βασικά χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης στρατηγικής που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τη διάσταση της ασφάλειας, αλλά και τις πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης, ασύλου, ανάπτυξης και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια άλλη πτυχή αφορά την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική διάσταση της ασφάλειας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που ασχολούνται σε θέματα δικαιοσύνη ιστορικών υποθέσεων θα πρέπει να δραματίσουν το ρόλο τους, στηρώντας πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουν αντίκτυπο στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας στην ε, στρατηγική εξωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις ε, που απορρέουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα των θεωρών να να πω η δικαιοσύνη, η δικαστική συνεργασία θα πρέπει να είναι θεμελιώδης διάσταση στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Παρά τα αυτά, αυτή η διάσταση έχει μόνο περιθωριακό χαρακτήρα στην πρώτη επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να ισχυθεί ε, η αστυνομική η δικαστική συνεργασία μεταξύ των μελών και η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να καταστήσει κοινωνού όλε τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών και του ευρωπαϊκού αρμόδιου οργανισμού. Χρειάζεται λοιπόν όλοι να εξετάσουν αυτή τη συνεργασία ω συνεργασία προτεραιότητα. Εντάχει, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τη έκθεση. Περιμένω βεβαίως και τις δικές σας προτάσεις, όπως και τις τροπολογίες σας και σας ευχαριστώ ε, εκ των προτέρων συνεργασία σας. Το μήνυμά μας είναι σαφές η πολιτική ασφαλείας δεν μπορεί να καταλήξει σε κάτι καθαρά επιχειρησιακό και τεχνοκρατικό. Είναι κατά κύριο λόγο ένα θέμα πολιτικό και άρα χρειάζεται ισχυρή δημοκρατική συνιστόσα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο από τους Ευρωπαίους ε, συνομοθέτες και από τους εθνικούς νομοθέτες που έχουν μείνει στην άκρη στο παρόν. Το Ευρωκοινοβούλιο όπως και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να είναι σε θέση να ε, εκφράσουν την άποψή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα όπως αυτά που από τις συνθήκες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Εγώ ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να παρέμβει πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θέλετε να μας πείτε κάποια στοιχεία ίσως χρήσιμα για τη συζήτησή μας. Ο κύριος Νούνας Ελμέιδα και μετά θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Δύο-τρία σημεία. Καταρχάς, να συγχαρώ την κυρία Μπορσελίνο και να την ευχαριστήσω και την ίδια αλλά και την ομάδα της για την πολύ αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Κάποια σχόλια για το σημείο 6 αυτής της έκθεσης. Γενικώ η έκθεση ε, μας ικανοποιεί για το σημείο 6 τώρα, συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις ε, πληροφορίες που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε εντός του ε, ευρωπαϊκής πολιτικής, είτε στο ιστορικό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε στο ιστορικό της Γενικής Διεύθυνσης Home για να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση ό,τι αφορά την αξιολόγηση απειλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σημείο 8 Συμφωνούμε απόλυτα. Προσυπογράφουμε το ότι πρέπει να υπάρξει μια ετήσια έκθεση και μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την ιστορική ασφάλεια. Για το σημείο 10, ε, ίσως εκεί να δυσκολευτούμε να δεχτούμε το ότι οι ανθρωπογενείς καταστροφές δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε όλο αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Νομίζουμε ότι και οι ανθρωπογενείς ε, καταστροφές ε, είναι ε, δόλιες πολλές φορές ή εγκληματικές. Οπότε μια στενάρη πολιτική προστασία των κρίσιμων υποδομών μας θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της εσωτερικής ασφάλειας, της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια. Για το σημείο 12 δεν έχουμε πρόβλημα για τις περαιτέρω αναφορές που κάνει η συγγήτρια, αλλά θα θέλαμε να επικεντρωθούμε σε κάποια από τα σημεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Οπότε θα πρέπει όντω να δούμε κατά πόσο υπάρχει σκοπιμότητα. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών ή επιχειρησιακών εγκλημάτων. Τώρα, για το σημείο 16 και την ρίζοσπαστικοποίηση. Ε, το αναφέρει η η, ε, η συγκεντρία, αλλά θα πρέπει να, δούμε, να πούμε ότι ε, εδώ μιλούμε για οποιαδήποτε μορφή ριζοσπαστικοποίηση και όχι κάποια συγκεκριμένη. τώρα, για το θέμα της ασφάλειας και της ασφάλειας των συνόρων, συμφωνώ ότι δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας στα σύνορα, αλλά στα πλαίσια της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια βλέπουμε τα σύνορα ως ένα εργαλείο ασφάλειας, γιατί είναι ένα μέτρο ασφάλειας. Είναι ένα εργαλείο βεβαίως και για τον έλεγχο τη πολιτική της πολιτικής Αλλά αυτό δεν εμπίπτει κατά ανάγκη στην εσωτερική ασφάλεια. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, άλλο κεφάλαιο ε, του οπλοστασίου πολιτικών που έχουμε. Τώρα, όπως ξέρει το Κοινοβούλιο, βεβαίως θα ενημερώσουμε και την Eurojust και την Europol και θα γίνουν κάποιες αξιολογήσεις επιπτώσεων Φυσικά ο έλεγχος από πλευράς Κοινοβουλίου είναι ένα από τα βασικά σημεία της ε, μεταρρύθμισης και πάλι όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπορσελίνο και την ομάδα της γιατί μας έφτασαν μέχρι εδώ και πραγματικά προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έξι έχουν ζητήσει το λόγο. 7. Η κυρία Χάγκης και αν θέλετε να προλάβουμε και το πρόγραμμα να είσαστε σύντομοι παρακαλώ. Μάλιστα πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πριν μιλήσω για την έκθεση της κυρίας Μπορσελίνο να πω δύο πράγματα για την πρώτη ετήσια έκθεση της Κομισιόν η οποία θεωρώ ότι αποτελεί μια πάρα πολύ καλή έκθεση επαγγελματική, εύληπτη για την κατάσταση ώστε να έχουμε μια εις άποψη για το τι γίνεται. Πρώτον λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Αλμέιδα και την ομάδα του που προετοίμασαν αυτό το πολύ καλό έγγραφο. Δεύτερον, η έκθεση της κυρίας Μπορσελίνο επίσης είναι εύληπτη και πολύ ισορροπημένη. Εκτιμώ πραγματικά την προσπάθεια που έκανε και θα ήθελα να της αναφέρω τα συγχαρητήριά μου. Με τα περισσότερα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει συμφωνώ. Για παράδειγμα, συμφωνώ απολύτως με τη συμφωνία που υπάρχει ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών, για την συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη και τις ε, υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο επίσης η ύπαρξη κοινών προτύπων για την αξιολόγηση των απειλών. Επίσης, πολύ σημαντικό, και εδώ συμφωνώ με την εισηγήτρια, είναι η σύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό ε, ε, ε, η προτινόμενη αξιολόγηση για την εξωτερική διάσταση να δίνει ένα σαφές μήνυμα ότι μιλούμε για δύο διαφορετικές, για δύο μάλλον πτυχές της ασφάλειας οι οποίες δεν μπορούν να διαχωρίζονται όπως έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο. Επίσης, κάτι άλλο με το οποίο συμφωνώ είναι το σημείο για τη σημασία που έχει το οργανωμένο έγκλημα. Το έχουμε συζητήσει πολύ. Ένα ίσονο σημασία όμως σχόλιο, παρατήρηση που θα ήθελα να προσθεθεί, είναι η διαφθορά το έγκλημα των λευκών κολάρων όπως ε, το λέμε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και συνδέεται και με το ποινικό έγκλημα. Υπάρχει ε, ο όρος αυτός, το λευκό κολάρο σε πολλές ε, χώρες. Ε, πέραν αυτή της μικρής τροποποίηση δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ε, εντάξει, υποθέτω ότι σε αυτό το σημείο θα συμφωνήσουμε με κάποιο τρόπο με την εισηγήτρια δεν θέλω να καθυστερήσουμε όμως, άλλο δεν θα μακρηγορήσω. Θα πω απλώς ότι στο σημείο αυτό η έκθεση ξεκινά με τα εκτιμώντας και τα λαμβάνοντας υπόψη. Ε, γίνεται μια αναφορά σε, ένα, σε κάποια ε, έγγραφα αναφοράς με, τις, ε, με τα σχέδια δράσης και τις στρατηγικές όπως ας πούμε το σχέδιο για την, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η στρατηγική για τις ευρωπαϊκές πόλεις κτλ. Ε, τελειώνω, Πρόεδρε. Ε, πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια νέα εκδοχή του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της Τρομοκρατία. Αυτά δεν αναφέρονται. Ή λοιπόν θα, θα αυξήσουμε την λίστα αυτή για να βάλουμε όλα τα σχετικά έγγραφα ή θα την κάνουμε πιο σύντομη και θα πούμε δύο-τρία μονάχα. Και κλείνω. Ένα ακόμα πράγμα να πω. Ο κύριος Αλμέιδα νομίζω το είπε. Κυρία Χάκης μπορείτε να κλείσετε. Νομίζω ότι πολλές φορές ε, έχει ε, αποδειχθεί ότι ε, σε κάποιες περιπτώσεις η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανταποκριθεί. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε από το ΕΛΚ την έκθεσή της με αυτές τις μικρές προσθήκες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Συναδελφοί, σας παρακαλώ να είσαστε πιο σύντομοι, δύο, το πολύ τρία λεπτά, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε ποτέ. Έχουμε δέκα λεπτά για το υπόλοιπο αυτής της συζήτησης, σκεφτείτε. Έχουμε άλλους έξι που θέλουν να μιλήσουν και έχουμε και την εισηγήτρια που θέλει να απαντήσει. Μείνετε αν θέλετε στα δύο λεπτάκια για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Εντάξει, τα δέκα δευτερόλεπτα δεν είναι τρομερό, εν πάση περιπτώσει, αλλά ε, Δείξτε και εσείς μια κατανόηση. Η κυρία Αλφάνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Μπορσελίνο, γιατί από την πρώτη στιγμή ενέπλεξε όλους τους σκιώδες εισηγητές. Υποστηρίζω την έκθεση πλήρως και μάλιστα έδωσε έμφαση στη σημασία συνεργασίας δικαστικών και ερευνητικών αρχών. Σωστό αυτό. Επίσης μίλησε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το θεσμικό ρόλο στην πολιτική ασφάλειας. Μ' άρεσε η αναφορά που έκανε στο οργανωμένο έγκλημα και ε, θυμάστε και την έκθεση που υιοθετήσαμε στις 25 Οκτωβρίου στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αναφέρεται σωστά το θέμα. Δηλαδή, λέει ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα ε, στον αγώνα ε, κατά της ε, εγκληματικότητας εναντίον του περιβάλλοντος. Αυτή η μορφή εγκλήματος έχει καταστρεπτικές συνέπειες λόγω της οικονομικής κατάστασης και στη ζωή των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό Ευχαριστώ που ήσασταν και λακωνικοί, κυρία Αλφάνο. Κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την ε, κυρία Μπορσελίνο. Στο τέλος της έκθεσης της λέει ότι ε, πρέπει να ξανασκεφτούμε ίσως το γενικότερο πλαίσιο που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Μιλούμε για τις αρχές της ε, ισότητας και της μη διάκρισης, ε, αρχές δηλαδή πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ακόμα και όταν ε, ασχολούμαστε με την ε, πολιτική για την ασφάλεια. Εγώ ήμουνα μέλος ενός Περιφερειακού Συμβουλίου για 10 χρόνια και μιλούσαμε για την ασφάλεια στους δρόμους, για την εγκληματικότητα, και λέγαμε ότι παντού θα μπουν κάμερες για να, να μπορούμε να προλάβουμε, για να βελτιώσουμε την κατάσταση κτλ. Αλλά ε, αυτοί που ε, διώκονται ή τέλος πάντων ερευνώνται τα στοιχεία τους έστω και προληπτικά συνήθως είναι μετανάστες ε, και μετά καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν και δημιουργούνται υποψίες ε, υπάρχει λοιπόν η μεμονωμένη ε, ελευθερία υπάρχει και η συλλογική ελευθερία και αυτό θα πρέπει να είναι σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής για την, για την ασφάλεια λείπουν κάποια σημεία εδώ φοβούμε όμως ότι πάμε σε μια κατεύθυνση τη συλλογική ελευθερία, η οποία ναι, μεν είναι επιθυμητή, αλλά να μην καταπατήσουμε, να μην καταστατηγήσουμε την ατομική ελευθερία. Η εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να, να ε, ε, συνδυαστεί και με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τους α, ε, ε, κινδύνους που υπάρχουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι καθήκον των διπλωματικών μας υπηρεσιών. Ε, πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σωστά. Θα είμαι, θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε, ε, αλλά νομίζω ότι αυτά που γράφονται στην έκθεση αντίκειται στο, στο άρθρο 21 της Συνθήκης γιατί και η εξωτερική μας πολιτική επίσης βασίζεται στη θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε μεταξύ του τι συμβαίνει εντός της Ευρώπης και του τι συμβαίνει εκτός αυτής. Είναι περίεργο, παράξενο κυρία Πρόεδρε, που δεν μπορούμε να κρίνουμε επιπίας βάσεως και ποιες επιπίες βάσεως έγιναν οι αναλύσεις για την ασφάλεια. Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο αυτό να το αναλύσει η Κομισιόν. Και αν το αναλύσει θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Με απογοήτευσε σε κάποιο βαθμό πάντως η έκθεσή σας, το ομολογώ. Όμως αυτά που είπατε στην αρχική σας παρέμβαση με καθησύχασαν κάπως. Και σε ό,τι αφορά ε, τον περιορισμό των λέξεων, ξέρω πολύ καλά ότι έχουν ε, επιπτώσει στο, στο τελικό κείμενο, στο πώ φαίνεται. Θέλω να κάνω κάποιε ε, τηλεγραφικές παρατηρήσεις, Πρόεδρε, να μου επιτρέπετε. Και εγώ θεωρώ ότι η ισορροπία μεταξύ ασφάλεια και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όταν διαβάζουμε την έκθεση βλέπουμε ότι η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια περισσότερο και όχι στον άλλο τομέα όλες οι ζημίες των δημοσίων ελευθεριών σε κάποια κράτη-μέλη εν ονόματι της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ε, είναι πολλές. Και σε μερικά κράτη-μέλη τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Θα πρέπει να υπαγρυπτούμε λοιπόν. Επίσης ξέρουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τη βία είναι η πρόληψη. Και νομίζω ότι και εδώ πρέπει να, βρούμε την, να ξαναβρούμε την ισορροπία. Γιατί σε αυτή την περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης ξέρουμε ότι πάντα αυξάνονται τα φαινόμενα βίας και επομένως ε, πρέπει να επαγρυπνούμε, χωρίς όμως να κάνουμε λάθος ούτε για τα μέσα, ούτε για τους πόρους που χρειαζόμαστε για να το πετύχουμε αυτό. Έχω ερωτηματικά για την ισορροπία, επίσης, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και του σεβασμού της επικουρικότητας. Στην ομάδα μου μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος ο σεβασμός αρχής επικουρικότητας, αλλά αυτό δεν είναι τέχνασμα για να απαλλάξουμε ορισμένα κράτη-μέλη ε, σε σχέση με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή απέναντι στην ε, σύμβαση, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που όλοι έχουν υπογράψει μία προς μία όλες οι χώρες. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε η Judith Σαρτζεντίνη Τελείωσα, Πρόεδρε, κυρία Ιντβελ. 30 δευτερόλεπτα δώστε μου. Η σχέση εσωτερικού και εξωτερικού παράγοντα, πούμε, και άξονα πρέπει να το ξαναδούμε, πρέπει να το ξαναδουλέψουμε αυτό το σκέλος. Επίσης, η ανάλυση των απειλών που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Κύρια Βερζιά, έχω άλλους τέσσερις ομιλητές. Σας παρακαλώ, καταλήξτε επιτέλους. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που μου, με εκνευρίζουν, ε, γιατί είναι πολύ αόριστες. Η απειλή ή ριζοσπαστικοποίηση. Αλλά θα κάνω και προτάσεις επ' αυτών. Ο κύριος Σάλβαρο, η κυρία Λάντφορντ και ο κύριος Σλούτερ και μετά η, η συγκέντρια. Ο κύριος Σάλβαρο, ευχαριστώ. Um, I also thank our colleague, Mrs. Να ευχαριστήσω την κυρία Μπορσελίνο για τη δουλειά που έκανε αλλά νομίζω ότι ε, υποτίμησε τις δυνατότητές της για το τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της ασφάλειας. Ε, ακόμα πολλά μπορούμε να κάνουμε και όπως είπε και ο κύριος Αλμέιδα προφανώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Ένα σημείο λοιπόν που δεν βλέπω στην έκθεση και νομίζω ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί είναι το πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλους οργανισμούς που ε, ασχολούνται με το θέμα της ασφάλειας όπως το ΝΑΤΟ, όπως ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, ο ΑΣΕ. Μπορούμε λοιπόν να επωφεληθούμε πολύ από την συνεργασία με άλλους οργανισμούς από ό,τι τώρα. Και επίσης κάτι άλλο που λείπει είναι το τι σημαίνει ασφάλεια. Έχουμε κάποιον ορισμό συγκεκριμένο για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η ασφάλεια. Μιλούμε για δημόσια ασφάλεια, ασφάλεια κρατών, το, το υποκείμενο της ασφάλειας. Τι ακριβώς σημαίνει ασφάλεια. Να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται όταν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Και όσο σημαντικό είναι να τονίσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικοί είμαστε όλοι, ε, εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια σε αυτούς τους διαφορετικούς τομείς. Οπότε, αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στην έκθεση και δυστυχώ δεν ξέρω πού να το βρω, η Κομισιόν δεν μας το έχει παρουσιάσει ποτέ, είναι ένα έτσι οργανόγραμμα ε, μιας νομοθεσίας που να υπάρχει στην τομέα τη ασφάλειας. Πώς συνδέεται, πώς δημιουργείται, πώ συνδυάζονται οι διάφορες νομοθετικές πράξεις, τι θα μπορούσε να γίνει στι προτάσει, σε ποια πρόταση θα μπορούσαν να εισαχθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Αν δούμε δηλαδή πω συνδέονται οι διάφορες ε, νομοθεσίες για την, για την ιδιωτικότητα των δεδομένων, για την προστασία των δεδομένων κτλ. Ξέρω ότι λιώνει και ο χρόνο μου. Οπότε, ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλή αρχή η έκθεση τη κυρίας Μπορσελίνο, αλλά πρέπει να τη βελτιώσουμε αν θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε όταν ε, μιλούμε για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η Βαρόνι Λάτφορντ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νούνες Δελμέιδα. Στην παράγραφο 10 η εισηγήτρια ε, απορρίπτει την ιδέα που λέει ότι οι καταστροφές και οι κρίσεις συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό των απειλών στην εσωτερική ασφάλεια ή την εξωτερική ασφάλεια. Νομίζω ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν, η αρχική ανακοίνωση της Κομισιόν, ε, δεν μιλάει μόνο για ανθρωπογενείς καταστροφές, αλλά και για φυσιολογικές καταστροφές ή κινδύνους. Όταν ας πούμε δούμε τι έγινε πέρσι στην Ιαβωνία, τσουνάμι, μετά η πυρηνική ε, καταστροφή και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν, μιλάμε για τις τηλεπικοινωνίες που καταστράφηκαν, την ενέργεια, τις μεταφορές, το ίντερνετ. Στην αρχική ανακοίνωση της Κομισιόν αυτό έμπαινε στο, στον γενικό τομέα της ανοχής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ή της αντίστασης. Ε, και το είπε και ο συνάδελφος Άλβαρο. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, με τη ΣΥΠΑ καταρχάς, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο σύνδεσμος που έχουμε, ο υπερατλαντικός. Οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται γιατί βεβαίω ε, πρέπει να συμπεριλάβουμε και το κυβερνό αλλά εδώ μιλούμε για πολύ πιο ευρεία πράγματα. Μέχρι το τέλος του 2012 η Κομισιόν θέλει να υποβάλει ε, μία έκθεση για, την, για τις ανθρωπογενείς καταστροφές και μετά θέλει μέχρι το 2014 να έχει ε, την, ε, ένα, ένα σύστημα αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών και των καταστροφών. Ε, όταν όμω έγινε κάποια στιγμή μια διακοπή των τηλεπικοινωνιών, εγώ δεν μπορούσα να έχω ίντερνετ από το τηλέφωνό μου. Καταλαβαίνετε πόσο εξαρτημένοι είμαστε. Α, τα αυτοκίνητά μα δεν λειτουργούν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα τη ασφάλεια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο τελευταίο των συναδέλφων, ο κύριο Σλούτερ από τη Σουηδία. Εν τω μεταξύ θέλει να παρέμβει και η Προεδρία του Συμβουλίου Παρακαλώ σύντομα στα δανέζικα όταν μιλήσετε. Ο κύριος Λούτερ, ήρθα εδώ στην ε, Επιτροπή ως αναπληρωματικό μέλος από την ΙΝΤΑ. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Μου αρέσει πάρα πολύ η παράγραφος 12 γιατί νομίζω ότι το έγκλημα κατά του περιβάλλοντος απειλεί την ασφαλειά μας ή τα τοξικά απόβλητα που απειλούν την υγεία μας, το ίδιο με την φτώχεια η φτώχεια. Αν είναι κάποιο ε, ε, πολύ φτωχό, προφανώ δεν θα τρέφεται καλά. Αν δεν τρέφεται καλά, δεν θα αναπτυχθεί σωστά. Όλα αυτά είναι απειλή για τη ζωή του. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα είναι ένα σημαντικό κομμάτι τη όλη στρατηγική. Και δεν θα ήθελα να μιλήσουμε τόσο πολύ για την ασφάλεια, αλλά για την ε, πολιτική άμυνα. Εντάξει, τώρα η εκφράση που χρησιμοποιώ μπορεί να είναι διαφορετική σε άλλε χώρε, αλλά ο κίνδυνο μια φυσική καταστροφή δεν είναι τόσο σημαντικός όσο ε, το πρόβλημα ή η απειλή για την, ε, για την υγεία. Και βλέπετε ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται τρομοκράτες για να καταστρέψουν τα δίκτυά μας. Μια βροχή αρκεί. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστή αντίσταση για όλα αυτά. Βεβαίω, εγώ δεν θα δεχτώ κανένα άλλο αντιτρομοκρατικό μέτρο εκτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν κάνει ε, οποιοδήποτε, μια μεγάλη ευρεία ανάλυση για την αποτελεσματικότητα, για το κόστο και για το κατά πόσο ε, επηρεάζονται τα θεμελιώδη μα δικαιώματα. Αν δεν την κάνει αυτή την ε, ανάλυση η Κομισιόν, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κανένα άλλο αντιτρομοκρατικό μέτρο. Οπότε ας αξιολογήσουμε παρακαλώ όλα τα δεδομένα. Φυσικά και μη. Ε, ευχαριστώ. Δεν, η, ο εκπρόσωπο τη Ελληνική Προεδρία δεν ξέρω το όνομά σα. Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο δανό και όσο σύντομο μπορώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ εκ μέρου τη ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ την κυρία Μπορσελίνο για την έκθεσή τη. Νομίζω ότι. Ε, είναι σημαντικά τα θέματα που θέτει και το ενδιαφέρον που δείχνει το Κοινοβούλιο σε όλα αυτά. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις απόψεις, ας πούμε. Βλέπω στο κείμενο ότι ζητείται μια συνολική ε, ανάλυση με βάση τον, ε, τον ε, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και τις αποδείξεις ε, για τις απειλές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το κάνει η Κομισιόν ε, και για πρώτη φορά γίνεται. Αυτό το σημείο ακριβώς ε, έχει να κάνει με την συμβολή στους νομοθέτες, με την παροχή πληροφοριών, έτσι ώστε να μπορούν να νομοθετήσουν. Επίσης, το αίτημα που υπάρχει για την αξιολόγηση του κύκλου των πολιτικών είναι αποτελεί ένα στόχο για το 2013. Και σε ό,τι αφορά την αναφορά που γίνεται ή το αίτημα που υπάρχει για πιο στενή συνεργασία εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της ε, ασφάλειας και της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το δουλεύουμε. Υπάρχουν πολλέ ε, επιτροπέ και στο Συμβούλιο Ομάδα Εργασία οι οποίε ασχολούνται με το θέμα τη ασφάλεια. Οπότε έχουμε προχωρήσει αρκετά και νομίζω ότι πάμε καλά. Επίση, υπάρχουν ε, κάποια σημεία με τα οποία δεν θα συμφωνούσαμε απόλυτα. Γιατί η εσωτερική ασφάλεια είναι πολύ ευαίσθητο τομέα. Και γι' αυτό μερικώ έχει αφαιθεί και στη δικαιοδοσία των κρατών μελών ειδικά όταν μιλούμε για την ιστορική ασφάλεια των κρατών μελών. Όταν βλέπουμε λοιπόν την αναφορά στην ε, συμπερίληψη στη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον όλο, στην όλη εικόνα πολιτική για το μέλλον, αυτό βεβαίω είναι ευαίσθητο θέμα. Όπω ξέρετε, Δίνω πληροφορίες στο Κοινοβουλίο για τη δουλειά που γίνεται ανεξάμεινο. Αυτά από μένα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ωραία. Τηρήσατε και το χρόνο. Κυρία Μπορσελίνο, θέλετε να απαντήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν, το Συμβούλιο, του συναδέλφου που πήραν το λόγο που γενικά ήταν ευνοϊκή απέναντι στην εκθεσή μου. Σίγουρα υπήρχαν ελλείψεις, αλλά οφείλονται κυρίως στις δυσκολίες του να πω πολλά με λίγες λέξεις. Θέλω να συμπληρώσω και να βελτιώσω το συντομότερο δυνατόν το κείμενο με την παρουσίαση τροπολογιών. Οι τροπολογίες και ε, των συναδέλφων, έτσι, όχι μόνο δικές μου, Χάρη σε επισημάσεις που έγιναν σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις, ε, θα έχω την ευκαιρία να διορθώσω. Ε, το θέμα είναι τόσο ευρύ, τόσο περίπλοκο, τόσο πλήρες. Υπάρχουν πολλά θέματα τόσο ευαίσθητα και λεπτά που πρέπει να τονιστούν με προσοχή. Για το ρόλο του Κοινοβουλίου, για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Αυτά είναι θέματα προτεραιότητας και εκ των όνου κάνευ για μας. Και θα τα αναφέρουμε και στην έκθεσή μας, το δίχως άλλο. Περιμένω λοιπόν συνεισφορές για να βελτιώσω το κείμενο και να το κάνω σαν τον πιο ικανοποιητικό, αποτελεσματικό κτλ. Υπενθυμίζω στους αδέλφους ότι σε 7 Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Και πάμε τώρα στο επόμενο σημείο, η σημεία μάλλον της μερικής διάταξης. Όλα σχετίζονται με τις διαδικασίες απαλλαγής. Έχουμε νέα εκθέσεις και 45 λεπτά για να τις εκπαιρεώσουμε. Είναι η έκθεση για την απαλλαγή για το 2010, για την Κομισιόν, το EDPS ε, και τις έξι, τους έξι οργανισμούς για τα θεμελιώδη δικαιώματα, Frontex, Europol, Eurojust, C-Pol την Αστυνομική Ακαδημία δηλαδή, και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθηση ε, Ναρκωτικών και Τοξικομανία. Και, το... και βεβαίως ε, για τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασία των Δεδομένων. Δεύτερο είναι αυτό. Έχουμε πέντε διαφορετικούς εισηγητές. Ορισμένοι έχουν ε, όχι μόνο μία εκθέσεις, αλλά παραπάνω. Άλλοι έχουν μόνο μία. Θέλω να δώσουμε το λόγο καταρχάς στους πέντε εισηγητές. Σύντομα παρακαλώ, πολύ σύντομα. Όσοι φεύγουν από την αίθουσα να φύγουν με πειθαρχία και ησυχία. Παρακαλώ, κάντε κάποια εισαγωγικά σχόλια για δύο ή τρία λεφτά. Γιατί θα χρειαστούμε ακόμα και έτσι 15 λεφτά και θέλω να αφήσω λίγο χρόνο για συζήτηση. Εν συνεχεία θα επανέλθετε με τις καταληκτικές σας παρατηρήσεις. Ο κύριος Φάντεν Κάμπα, ο κύριος Μπουσουτήλ, Σάμερ, Ματιέ και Γιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνο για δύο εκθέσεις, όπως είπατε κι εσείς. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία με το προσωπικό και τη συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού ε, για θέματα που αφορούν κυρίως ε, την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Γενικά το 2010 η κατάσταση ήταν καλή. Οι οργανισμοί ε, εξόδεψαν σωστά τα κονδύλια τους Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις βέβαια, επικριτικές που ανέφερα στην εκθεσή μου. Υπάρχει μια υποεκμετάλλευση των οικονομικών μέσων από κάποιους οργανισμούς και όταν υπάρχει δημοσιονομική λιτότητα σε εθνικό επίπεδο, το να, ζητάνε, να ζητάμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περισσότερα λεφτά τα οποία δεν απορροφώνται εν συνεχεία, αυτό είναι αδικαιολόγητο. Εδώ συζητάμε τα προγράμματα εργασίας, τα ετήσια προγράμματα. Αλλά τι νόημα έχει να τα συζητάμε αν δεν υπάρχει απορρόφηση των πόρων. Κάνουμε λοιπόν κάποιες προτάσει για κάποιους οργανισμούς και τους λέω προσοχή ε, στο πω ξοδεύετε τα λεφτά. Με συνεχεία, για το προσωπικό. Δεν έχουν ε, πληρωθεί όλες οι θέσεις ακόμα. Υπάρχει ο προπολογισμό όμως. Εμείς ούτως ή άλλως, ε, εμείς ως Κοινοβούλιο πήραμε την απόφαση να υπάρξουν αυτές να πληρωθούν αυτές τις θέσεις, οπότε είναι κατανόητο γιατί δεν έχει γίνει. Τώρα, ε, υπάρχει μια μείωση των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων και αυτό δεν είναι σωστό για τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Για τη ΣΕΠΟΛ, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Με την κυρία Ματιέ για την περσινή απαλλαγή το, του 2009 το είχαμε συζητήσει και είχαμε εντοπίσει το ίδιο πρόβλημα. Τώρα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ ΣΕΠΟΛ και Europol. Ελπίζω η κατάσταση να βελτιωθεί για τη ΣΕΠΟΛ. Αυτά σταματώ εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ήδη σας υπερψήφισε κάποιος ε, από το Λαϊκό Κόμμα. Έχει καλή διάθεση. Τον βλέπω. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Έχω συντάξει την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Επόπτη, για το Frontex και για την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, για αυτές τις τρεις υπηρεσίες το ελεγκτικό συνέδριο έχει καταλήξει ότι οι πληρωμές για το 2010 ήταν σύμμορφες με τους κανόνες και ε, με βάση το σύστημα ελέγχου. Θέλω να κάνω κάποιες ε, επικρίσεις παρόλα αυτά. Λέω ευθύ εξ αρχή ότι το συμπέρασμα είναι θετικό. Προτείνω δηλαδή να χορηγήσουμε την απαλλαγή στι τρει αυτέ υπηρεσίε, στου τρει αυτού οργανισμού. Για τον Ευρωπαίο Πόπτη Προστασία Δεδομένων, καταρχά, η Ε, ο εσωτερικό διαγωνισμό σε τέσσερι διαφορετικού τομεί ε, οργανώθηκε από τον οργανισμό το 2009. Και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η οργάνωση όπως σας είπα, ενό εσωτερικού διαγωνισμού στον οργανισμό αυτό. Δεν άνοιξε ο διαγωνισμός ε, όπως γίνεται συνήθως μέσω της διαδικασίας έψω. Η DPS, ε, για να το δικαιολογήσει, είπε ότι ήταν ειδικά πόστα, ειδικέ θέσεις. δεν νομίζω ότι είναι καλή δικαιολογία αυτή, γιατί αυτό σημαίνει ότι κανένα εξωτερικός ε, που δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή ήδη το γραφείο αυτό η DPS δεν μπορεί να, κάνει, να υποβάλει τα χαρτιά του για αυτά τα πόστα. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε στην DPS ότι οι διαγωνισμοί έψω, οι κλασικοί διαγωνισμοί όπως τους ξέρουμε, είναι κατά πολύ καλύτεροι και επιθυμητοί. Σε ό,τι αφορά την ε, Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το ελεγκτικό συνέδριο κατέληξε στο πόρισμα ότι ακόμα μια φορά υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο δαπανών στο τέλος της χρονιάς. Φανταστείτε ότι αυτή η υπηρεσία ξόδεψε σχεδόν το μισό του προπολογισμού της το Δεκέμβριο. Δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά. Δεν είναι σωστό αυτό και θα πρέπει να τους επιστήσουμε την προσοχή να μην το ξανακάνουν, γιατί το έχουν ξανακάνει. Υπάρχουν επίσης κάποιες δυσκολίες ε, με την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την πρόσληψη, τη διαδικασία προσλήψεων, ένα σημείο που έχει ήδη τεθεί και ξανασυζητηθεί και μόνο 59 από τις 72 θέσεις πληρώθηκαν μέσα στο 2010, το οποίο δεν είναι σύμμορφο με τις απαιτήσει που μας λέει η υπηρεσία, που μας λέει ότι έχει υπηρεσία, ότι θέλει περισσότερες θέσεις και όμως δίνουμε τις θέσεις και μετά δεν τις καλύπτει. Αυτή η παρατήρηση δεν ισχύει μόνο για το 2010, την κάνουμε και πέρυσι για το 2009. Άσε Όπως και πριν, όπως είπα και πριν, καλό θα ήταν να μην ξαναδούμε να επαναλαμβάνεται αυτή η κατάσταση και του χρόνου. Το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα τώρα. Τέλος, σε σχέση με τη Frontex. Το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι μεταφέρονται πολλά κονδύλια από τη μια χρονιά στην άλλη. Η υπηρεσία αυτή μας λέει ότι υπάρχει μια απρόβλεπτη φύση στις δικές της αποστολές. Δεν ξέρει πότε θα αναγκαστεί να οργανώσει μια αποστολή. Σωστό αυτό. Γι' αυτό ακριβώς έχει τόσα μεγάλα ποσά μεταφοράς, που μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά δηλαδή. Ε, Εντάξει, το δεχόμαστε αυτό. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι ο προπολογισμό του οργανισμού πρέπει και μπορεί να προβλέπεται ε, και να οργανώνεται και να ετοιμάστε με έναν τρόπο που να μην γίνονται τόσε μεταφορές. Με τη νέα εντολή θα έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες η υπηρεσία και θα έχει πολύ περισσότερο προσωπικό και θα αναγκάσει να ξοδεύει πολύ περισσότερα χρήματα. Πρέπει παρόλα αυτά κατά την άποψή μου, να δώσουμε την απαλλαγή ε, σε αυτές τις τρεις ε, υπηρεσίες και να, πούμε, να συστήσουμε δηλαδή θετική, να πούμε ότι έχουμε θετική γνώμη στην ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για αυτές τις απαλλαγές. Ζόμερ. Ευχαριστώ για την απαλλαγή της Europol και της Eurojust. Καταρχάς για την Europol που δεν προέκυψε καθόλου. Ο προπολογισμό αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση για το 2010 και όλα τα, τις βασικές ε, συναλλαγές, όλες ε, τηρούν τις ε, προϋποθέσεις. Κυρίως μιλούμε για κάποιες μεταφορές από, την, από το ένα άτομο στο άλλο σε σχέση με τα κόστη. Η Europol έκανε και μετακόμιση στα νέα κεντρικά της γραφεία, οπότε καταλαβαίνετε για το έξοδο τι ακριβώς σημαίνει. Τώρα για τα μέτρα θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα ώστε να μειωθούν αυτές οι μεταφορές ε, ε, ποσών από το ένα έτος στο άλλο. Για το 2012 η καταγραφή του προπολογισμού θα πρέπει να ελέγχεται ε, μηνιαίως, κυρίως για αυτές τις μεταφορές ποσών. Αν μπορέσουμε αυτά να τα τηρήσουμε, υποθέτω ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις ροές πληρωμών. Οπότε συμφωνούμε και προτείνω να γίνει η απαλλαγή. Επόμενο σημείο για τη Eurojust. Εδώ το αιτήσιο συλλογισμό στα ουσιώδη του σημεία αντικατοπτρίζει την κατάσταση του 2010 και βεβαίως όλες οι α, συναλλαγές έγιναν νομίμως και σύμφωνα με το τυπικό, αλλά υπήρξαν κάποια έξοδα πολύ ψηλά το 2010 12 ε, η αιτιολογία είναι ότι υπήρξαν κάποια, προ, έτσι, κάποια υποδομές που αγοράστηκαν καινούργια κομπιούτερ για την, και δημιουργήθηκε το σύστημα για την διαχείριση των δεδομένων. Ε, καλό είναι ότι υπάρχουν ε, ήδη μέτρα που έχουν προβλεφθεί για το 2012 για την καθεοντότητα και για τα, κόστη, για τα έξοδα που κάνει και οι δεσμεύσει ό,τι αφορά την κατανομή των συμβάσεων θα πρέπει να γίνονται ε, το συντομότερο δυνατόν. Βεβαίως θα πρέπει να τηρηθούν όσα έχει ε, προβλέψει η υπηρεσία και θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Επίσης υπάρχει άλλο ένα σημείο που θα πρέπει να διορθωθεί ότι ο διχειριστικός διευθυντής δεν είναι υπεύθυνο για το καθημερινό και την καθημερινή διαχείριση ε, του κολεγίου που θα έπρεπε να είναι. Η Eurojust ε, θα πρέπει να λύσει το θέμα αυτό, να το εξετάσει το συντομότερο δυνατόν και αν εξακολουθήσουν να υπάρξουν ασυνέπειες και ασάφειες στο σημείο αυτό, ο νέος κανονισμός για τη Eurojust θα πρέπει να τις, ε, να τις μελετήσει και να τις άρει. Δεν τηρήθηκε σε ό,τι αφορά την, τα όσα λέει η Επιτροπή εξολογηση οι προβλέψεις που είχαν υπάρξει, η Γιώργος όμως λέει ως απάντηση ε, ότι ο, διαχειριστ, ο διευθυντής έχει, θα λάβει μάλλον ένα ευρύ λεπτομερές έγγραφο που θα μιλά για όλες τις συμβάσεις που δόθηκαν στην ε, περίοδο αυτή. Η Eurojust ε, λέει ότι θα ε, συνάπτει τις συμβάσεις αυτές νομίμως κτλ. και ότι θα, τηρήσει την, θα ενισχύσει μάλλον την αξιοπιστία της υπηρεσίας. Και ένα τελευταίο σημείο κριτικής. Υπάρχει για μια παλιά λίστα αναμονής η Eurojust θα πρέπει να δει την ισχύ αυτών των ληστών αναμονής που υπάρχει, ώστε να μην υπάρξει παρόμοια περίπτωση στο μέλλον. Η Eurojust μας είπε ότι όταν γίνονται κάποιες αναστολές με βάση αυτή την ε, λίστα αναμονής, ε, γίνονται μόνο σε μεμονωμένε ε, περιπτώσεις. Θετικό είναι ότι θέσεις εργασίας από 24% το 9 πήγανε σε 13% το 2010. Βεβαίως αυτό δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό όπως είπε και ο συνάδελφος Φάντερ Κάμπ. Ούτως ή άλλως ο προπολογισμός υπάρχει για τις θέσεις, οπότε οι θέσεις αυτές θα πρέπει να, να πληρωθούν. Οπότε δεν θα πρέπει να δαπανώνται χρήματα για θέσει που δεν ε, καλύπτονται. Οπότε προτείνω να συμφωνήσουμε για την απαλλαγή για την Eurojust. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ιντβελτ που με αντικαταστήσατε σε αυτό το πρώτο τμήμα συζήτηση ε, για τα θέματα των απαλλαγών. Κυρία Ματιό, νομίζω για την απαλλαγή του 2010 για το ΣΕΠΟΛ. Το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι πάνω από 1,6 δις ευρώ είναι μεταφορές από το 2009. Και αυτό είναι αντίθετο προς την δημοσιονομική αρχή της, του ετήσιου χαρακτήρα. Επίσης, η διαδικασία που χρησιμοποιεί το Σώμα των Επιτρόπων για να εγκρίνει την ε, δήλωση για, τα, για τις δαπάνες ε, δεν είναι ε, δεν έχει τη δέουσα αυστηρότητα σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά έγγραφα κυρίω. Δείχνει μια χαλαρότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και, υπάρχουν κάποια καλά νέα για τη ΣΕΠΟΛ. Σε ό,τι αφορά τι διαφορετικέ αλλαγέ τη οργάνωση τη υπηρεσία, με ικανοποίηση σημειώνουμε την απόφαση του Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου που καταργεί κάποιε επιτροπέ στο εσωτερικό τη Υπηρεσία αυτή. Η απόφαση που δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Σώμα ε, αστυνομία λέει ότι το Δημοδουσού μπορεί να δημιουργήσει ομάδε εργασία για λόγου συμβουλευτικού κους όταν υπάρχει ανάγκη και η ΣΕΠΟΛ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012 είχε άπειρες ομάδες εργασίες, επιτροπές, υποεπιτροπές κτλ. Και μετά από την πενταετή ετήσια έκθεση νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάποιος εξορθολογισμός οργάνωσης της ΕΠΟΛ ε, ούτως ώστε να μην έχουμε επικαλύψεις. Είμαστε σε καλό δρόμο για αυτό το θέμα. Το ίδιο για την αποτελεσματικότητα. Ο διευθυντή μαζί με τη γραμματεία θα πρέπει να μπορεί να παίρνει κάποιε αποφάσει που αφορούν την οργάνωση, χωρί αυτέ οι, α... οι ίσονο σημασία αποφάσει να πρέπει να επικυρώνονται από το δουσού. Ε, χαιρετίζουμε λοιπόν τον αριθ... τη μείωση του αριθμού των ατόμων του δουσού που ήταν 54 το 2010 και πήγαν στα 34 το 2011. Το δουσού λοιπόν θα ασχοληθεί με τα καθήκοντα της ε, υπηρεσίας και ο διευθυντής θα ασχοληθεί με τη διαχείριση. Για την καλύτερη σχέση των συνεδριάσεων του Δουσού, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να πούμε ότι το ΣΕΠΟΛ ε, δέχεται την μία σύμβαση του Κοινοβουλίου, δηλαδή ε, όλο και λιγότερα μέλη του, της ΕΠΟΛ θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δουσού. Γυρνάμε μία σελίδα, γιατί έχει απίστευτο παρελθόν αυτή η υπηρεσία. Ε, είχαμε κάποια κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για ιδιωτικούς λόγους. Ε, ανακτήσαμε κάποια χρεωστήτως καταβληθέντα στον από τον προηγούμενο ε, διευθυντή. Βρήκαμε λοιπόν κάποια κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακολίνο. Για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κέντρου ναρκωτικών και τοξικομανίας. Πολύ σύντομα. Ασχολήθηκα με την απαλλαγή του παρατηρητηρίου ε, για το 2010 που εδρεύει στην Λισαβόνα και που ασχολείται με την τοξικομανία. Έχω διατυπώσει κάποια ερωτήματα ε, που θα πρέπει να απαντήσει ο διευθυντής κ. Γκότς. Ε, μου απάντησε, είναι ικανοποιητικέ το ίδιο αποτέλεσμα, περιμένουμε μάλλον τα αποτελέσματα από το ελεκτικό συνέδριο. Τα οικονομικά είναι σε τάξη. Το παρατηρητήριο θα πρέπει να κάνει και επιπλέον προσπάθειες εξορθολογισμού των δαπανών, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, να υπάρχει ανταλλαγή καλών πρακτικών με τις υπόλοιπε ε, υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με τα ίδια θέματα σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ε, ένας, ε, μια ουσιαστική γραμμή του προπολογισμού για το Πρατήριο της Λισαβόνας στις επόμενες δημοσιονομικές, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο, μια νέα εντολή και χρειαζόμαστε μια στρατηγική που να μην αφορά μόνο την τοξικομανία αλλά και τις άλλες μορφές εξάρτησης το στίχημα στο ίντερνετ, την εξάρτηση από τον καπνό, το κάπνισμα κτλ. και άλλες εξαρτήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής. Εμείς δίνουμε θετικό, στέλνουμε θετικό μήνυμα και προτείνουμε να χορηγηθεί η απαλλαγή στην υπηρεσία αυτή. Κύριε Γιακολίνο. Ακούσαμε και τους πέντε εισηγητές για τα θέματα αυτά. Έχουμε νέα φακέλους απαλλαγών. Μπορούμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό, έχουμε λίγο χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που θέλουν να πάρουν τον λόγο. Η κυρία Ιντβέλτε. Yes, thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι Σκιώδης για την έκθεση Μπουστήλ για τον οργανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα πολύ σημαντικός οργανισμός ε, για μένα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι πολύ σημαντικό, άρα ο σχετικός οργανισμός θα πρέπει να έχει καλή λειτουργία. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, είπατε σχεδόν το ίμιση του προπολογισμού τελικά είχε δεσμευτεί μόνο για το τελευταίο μήνα του έτους και ρωτώ πώς ο οργανισμός μέσα τους προηγούμενους μήνες αρνήθηκε με αυτόν τον τρόπο να κάνει την έκθεση για τα μέσα ενημέρωση στην Ένωση. Αρχικά είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την έκθεση γιατί δεν έχουμε οικονομικούς πόρους και μετά δεν έχουμε εντολή. Δηλαδή πώς γίνεται να λένε ότι δεν έχουν πόρους και στο τέλος χρονιά να φαίνεται ότι υπάρχει ο μισός προπολογισμός. Ο δεύτερο ερώτημα, άλλης φύσεως. Ίσως είδατε στο διαδίκτυο ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο εξετάζει μια υπόθεση την οποία έφερε στο δικαστήριο ένα συνεργάτη του οργανισμού με την κατηγορία της παρενόχλησης. Στον λόγο άτομο ε, κατήγγειλε παρατυπίες πριν από μια διετία, τις οποίες χαρακτηρίζει παρενόχληση από τον επικεφαλής του οργανισμού. Εδώ βεβαίως δεν μιλούμε για την απαλλαγή του προπολογισμού, αλλά μιλούμε για την ποιότητα και τον ε, και τη συμπεριφορά του προσωπικού. Ε, έχουν υπάρξει τέτοιου είδου παρατυπίε στη συμπεριφορά του προσωπικού και έχουν επιληθεί έκτοτε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ινβελτ. Κυρία Ρονκέλα. Ευχαριστώ. Ε, εγώ είμαι σκιώδης για όλες τις εκθέσεις απαλλαγής. Ευχαριστώ όλους για τις εκθέσεις, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτές γιατί τα πλέον σημαντικά σημεία είναι μέσα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο εκτός βεβαίως από το γεγονός ότι δεν με κατανοώ το επιχείρημα της Frontex ότι είναι δύσκολο να κάνει προβλέψη του προγραμματισμού αλλά γιατί η Europol ή κάποιος άλλος οργανισμός, το EDPS, ε, μπορούν να προγραμματίσουν πολύ καλύτερα προβλέποντας τις επιχειρήσεις που έχουν να αναλάβουν. Το κατανοώ μεν, αλλά δεν μπορούν να το θεωρήσουν μια δικαιολογία γιατί θα πρέπει να το χρησιμοποιούν όλοι. Για την ΣΕΠΟΛ, την Αστυνομική Ακαδημία, μια ακόμη χρονιά να μας απασχολεί η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Πάντως εγώ αν ήμουν επικεφαλής της ΣΕΠΟΛ, θα προσπαθήσω να διασφαλίσω μετά από μία αποτυχία να λάβουμε απαλλαγή, θα έπρεπε τελικά να δείξουμε το καλό παράδειγμα και να είμαστε πρωτοπόροι. Ναι, μεν έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις της ΕΠΟΛ, αλλά πολύ μικρής κλίμακας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πέρα από όλα αυτά, ίσως με κάποιες μικρές αλλαγές στις εκθέσεις, εγώ θεωρώ ότι οι εκθέσεις σας ήταν εξαιρετικές και σας συγχαίρω για αυτές. Ευχαριστώ.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 Uh, Για το δεύτερο σχόλιο δεν έχω καμία εγώ ιδιαίτερη πληροφόρηση, αλλά αν πραγματικά συμβαίνει κάτι σοβαρό, τότε ναι. Βεβαίω πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα και να περιμένουμε απαντήσει. Από ό,τι καταλαβαίνω όμω δεν είναι θέμα οικονομικό, δεν είναι θέμα δημοσιονομικό και αυτή τη στιγμή μιλούμε για την απαλλαγή από την εκτέλεση του προπολογισμού, δεν πρέπει να θέσουμε θέματα παρενόχλησης προσωπικού. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά αν ε, θέλετε να κάνουμε μια εξέταση και έναν έλεγχο τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, εγώ θα σε υποστηρίσω. Πρόεδρος, θέλει κανείς άλλο το λόγο, έχει στήσει κανείς άλλο το λόγο ή κάποιος άλλος εισηγητής που θέλει να τοποθετηθεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να υπογραμμίσω κάτι για τις ε, θέσεις που δεν έχουν ε, πληρωθεί. Ε, το είπε και ο συνάδελφος. Σε σχέση με την Eurojust. Νομίζω ότι γενικώ θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Τι γίνεται με τις υπηρεσίες μας. Οι υπηρεσίες πάντα λένε ότι τους κατηγορούν ότι καταχρώνται, όχι καταχρώνται, ότι εν πάση χρησιμοποιούν πολλά χρήματα ενώ δεν τα χρειάζονται. Απ' τη μία βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ναι υπάρχουν κάποιες άδειες θέσεις. Αυτό θα μπορούσε όντω να αποτελεί έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά ίσως να μπορούσε να ερμηνευθεί και το όσο ότι ε, αυτή στιγμή οι θέσεις αυτές ε, δεν ε, πληρώνονται, πάνω να πει ότι δεν χρειάζονται κιόλας. Οπότε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να τη δούμε πολύ προσεκτικά και, στα επόμενα, και για τα επόμενα χρόνια. Να σκεφτούμε δηλαδή αν όντω αυτέ οι θέσει χρειάζονται. Ίσως θα μπορούσε να είναι αυτό μια προειδοποίηση για όλε τι αντιπροσωπείε, όχι μόνο, για, για όλες τις υπηρεσίες, συγγνώμη, όχι μόνο για την Eurojust. κυρία να, απαντήσω και εγώ σε συνάδελφο για τη ΣΕΠΟΛ εγώ δεν μπορώ να κάνω το συνήγορο της ΕΠΟΛ, αλλά ο Διευθυντής ε, είναι ακόμη στη διαδικασία να ξαναφέρει στην τάξη τα ε, πράγματα στην ΣΕΠΟΛ. Σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, να πω ότι οι σχέση εκεί δεν είναι τόσο απλές και δεν πιστεύω ότι τα πράγματα διευκολύνει με τις στάσεις και η Επιτροπή. Πιστεύω ότι θα πρέπει σε Πολ να έχει την ευκαιρία να ε, μας δείξει τι ικανότητες έχει στο μέλλον. Ο κύριος Δικολίνη, ναι, ε, σε ό,τι αφορά το δικό μου θέμα δεν υπήρξαν σχόλια, οπότε επιβεβαιώνω εκ νέου αυτά που είπα στην πρώτη μου παρέμβαση. Πρόεδρος, ωραία. Άρα κλείνουμε τη συζήτηση και για τις νέα εκθέσεις απαλλαγής και να συνοψίσω προτείνοντας το εξής. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 31η Ιανουαρίου. Το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 9 Φεβρουαρίου. Καλώς τροπολογίες, επαναλαμβάνω, έως τις 31 Ιανουαρίου το μεσημέρι και υπενθύμηση. Επειδή ενημερώθηκα από τις υπηρεσίες μας, οι τροπολογίες μπορούν να, να υποβληθούν συγγνώμη, μόνο στα αγγλικά. Ναι, ναι, ναι, μόνο στα αγγλικά. Έτσι. Έτσι γίνεται για κάποιο λόγο. και θα πρέπει να υποβληθούν με τα template του Word υποχρεωτικά σε αυτό το μορφότυπο. Σε Word templates. Έτσι είναι θέμα λογισμικού. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμη πληροφορία να την έχετε υπόψη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Αν θέλετε διαμαρτυρηθείτε, διαμαρτυρηθείτε και εγώ θα διαβιβάσω τα σχόλιά σας. Όμως, Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να σας το πω. Κοιτάξτε τώρα. Έχουμε ακόμη ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη που αφορά τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για τη διαβίβαση και τη χρήση δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών, για δεδομένα PNR. Έχουμε μία έκθεση την οποία θα μας παρουσιάσει η κυρία Πρίμπερ, ο κύριος Πρίμπερ, ο οποίος όμως δεν έχει έρθει ακόμη. Λοιπόν, να κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα μέχρι να έρθει. Τον περιμένουμε. Από λεπτό σε λεπτό. Ας ξαποστάσουμε λοιπόν για λίγα λεπτά. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό το τελευταίο σημείο για σήμερα θα συντηθεί και κλεισμένον των θυρών. Άρα, ποιοι είναι οι κανόνες για τη συνεδριάση και κλεισμένων των θυρών. Στην αίθουσα παραμένουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν προκειμένου, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας της, του Κοινοβουλίου, του Γραφείου του Προέδρου, την Νομική Υπηρεσία και εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων. Όπως και εκπρόσωποι της Γραμματείας Επιτροπής Λίβε. Μόνο αυτοί μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα.